Sehr äh, Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην συνεδρίαση της ε, Νομικής Επιτροπής ε, σήμερα και αύριο. Προτού να προχωρήσουμε στο πρώτο θέμα της ημερησίας διάταξης, ε, θα ήθελα να καλωσορίσω τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και την ομάδα του, τον κύριο Σκουρί και τους συνεργάτες του. Επειδή τα αποτελέσματα της συνεδρίασης των ε, ε, συντονιστών ε, είναι πολλά, θα ήθελα να τα αναβάλουμε και να περάσουμε κατευθείαν στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Θα ήθελα να ανακοινώσω το εξής, ότι στο, 30, στο σημείο 30 της ημερησίας διάταξης θα συζητήσουμε τα εξής. Καταρχήν, την ε, συνεδρία των συντονιστών, ε, την οποία είπα ότι θα αναβάλουμε για μετά την ακρόαση, επειδή έχουμε πολλά θέματα εδώ. Ε, μετά το σημείο 12 της ημερησίας διάταξης, τα λέω στα αγγλικά, τροπολογίες για την ε, γνωμοδότηση για τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Θα συζητήσουμε αυτό ε, το θέμα, διότι πρέπει να ε, εργαστούμε γρήγορα, διότι η Επιτροπή ΕΚΟΝ ε, θα ψηφίσει τη δική της έκθεση. Μετά το σημείο 21 της ημερησίας διάταξης θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων για την έκθεση της κυρίας Μακάρτη για τη διαφάνεια και αμέσως μετά θα έχουμε την ψηφοφορία για την οδηγία ε, όπου είναι εισηγητή ο κύριο Λένε για την ε, υποβολή λογαριασμών. Αυτό συνδέεται με το θέμα της διαφάνειας. Μετά το 27 της ημερησίας διάταξης ε, θα ψηφίσουμε σχετικά με τη συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ρωσική Ομοσπονδία πάνω, στους, πάνω στις πρόδρομες ουσίες των ναρκωτικών. και εδώ υπεύθυνος είναι ο κύριος Ρόμπλο και θα ήθελα να ανακοινώσω επίσης ότι η νομική βάση, ε, η νομική βάση για την ε, ισότητα μεταξύ των φύλων ε, δεν θα συζητηθεί αυτή τη φορά, θα αναβληθεί. Δεν θα ψηφιστεί δηλαδή αύριο. Τέλος, θα ψηφίσουμε τις τροπολογίες για, τον, για, για τη φορολογία επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και είναι απαραίτητο εδώ και αποφάσισα να μην γνωμοδοτήσουμε με κλασική γνωμοδότηση όπως κάνουμε συνήθως, αλλά λόγω της πίεσης του χρόνου είναι απαραίτητο να υποβάλουμε κατευθείαν τις τροπολογίες μας στην ΕΚΟΝ, στο όνομα του κυρίου Λένε και στο δικό μου όνομα. Διότι αλλιώ λόγω τη πίεση του χρόνου δεν θα μπορούν να ληφθούν υπόψη οι τροπολογίε αυτέ. Τέλο, έχουμε το σημείο 23 στην ημερήσια διάταξη, την έκθεση του κυρίου Καρύμ. Αυτή ε, θα συζητηθεί μαζί με το σημείο 22 της ημερησίας διάταξης, ε, που είναι επίσης του κύριου Καρίμ. Αυτά τα δύο θέματα δηλαδή ε, της ημερησίας διάταξης θα ε, συζητηθούν ταυτόχρονα. δεν έχουμε ε, ανακοινώσει του Προέδρου. Προχωράμε λοιπόν γρήγορα. Φτάνουμε στο σημείο 3 της ημερησίας διάταξης, έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης τα έχετε μπροστά σας. Ε, είναι από τις 18-19 Μαρτίου του 2013. Εάν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση μπορούμε να ολοκληρώσουμε και αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Τα αποτελέσματα ε, της συνεδρίας των ε, συντονιστών, όπως σας είπα, θα τα συζητήσουμε αργότερα. Και έτσι φτάνουμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης, στην ακρόασή μας. Και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να ξανακαλωσορίσω θερμά τον ε, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, τον κύριο Σκουρί, ε, και να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Αλεξάνδρα Τέιν. Α, Όχι, ζητώ συγγνώμη. Ε, θα δώσω πρώτα τον λόγο στον κύριο Σκουρί, που είναι πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα κάνω την ε, παρουσίασή μου στα γαλλικά, που είναι η γλώσσα εργασία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Κυρίε και κύριοι, καταρχήν θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μου απευθύνατε να μιλήσω ενώπιόν σα ε, περί τη μεταρρύθμιση του ε, Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα σας παρουσιάσω καταρχήν τις πρώτες γενικές ε, γραμμές και μετά τα αποτελέσματα που έχουμε ε, ε, ήδη από μια μερική μεταρρύθμιση που έχει οθετηθεί μέχρι τώρα. Τέλος, θα σας μιλήσω για το θέμα της μεταρρύθμισης που δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί πριν κλείσω με κάποιες σκέψεις πιο γενικές. Η μεταρρύθμιση που πρότεινε το δικαστηρίο το Μάρτιο του 2011, πριν από πάνω από δύο χρόνια δηλαδή, προς τα νομοθετικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αφορά ε, τα τρία σώματα ε, που το απαρτίζουν. Η πρόταση αφορά τη μεταρρύθμιση των κανόνων της σύνθεσης, ε, της μίζωνος σύνθεσης, της λειτουργίας των Προέδρου και Αντιπροέδρων, την αύξηση των αριθμών των δικαστών και την δυνατότητα ε, ε, ε να ε, προσληφθούν ε, προσωρινοί δικαστές στα ειδικά τμήματα. Η απόφαση του Συμβουλίου του 2012 επέτρεψε κάποιες μεταρρυθμίσεις. Μετά την ανανέωση των μελών το 2012 εξελέγει ένας αντιπρόεδρος και άλλαξε η σύνθεση της μίζων, η μίζων ε, σύνθεση. Ε, απαρτίζεται από 15 αντί για 13 ε, δικαστές, πρόεδρο, αντιπρόεδρο, τρεις πρόεδρους τμήματων, πέντε δικαστές και άλλους δικαστές. Σε ό,τι αφορά για τους προσωρινούς ε, δικαστές του Δικαστηρίου Ευρω... ε, Δημόσιας Διοίκησης, Έχουμε ένα κανονισμό ε, και υιοθετήθηκε προχθές ε, η κατάλληλος που είχα προτείνει για τρεις προσωπικότητες οποίες θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε να καλέσουμε για να, να αντικαθιστούμε ένα δικαστήριο όταν αυτός αδυνατεί να εκπληρώσει τα καθήκοντά του. Σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση ε, που έχει υιοθετηθεί. Ήδη έχει δώσει καρπούς η συμμετοχή ενός μεγαλύτερου αριθμού δικαστών στην μείζωνα σύνθεση. Έγινε δυνατή και ασφαλώς ε, βελτιώνεται το κύρος των αποφάσεών της. Αλλά ακόμα πιο σημαντικό, η δημιουργία ενός, ε, μιας, ενός πέντου τμήματος πενταμελούς επέτρεψε να μπορούμε να εκδικάζουμε παράλληλα μεγαλύτερο ρυθμό υποθέσεων. Αυτή τη στιγμή έχουμε πέντε αντί για τέσσερα πενταμελή τμήματα. Ε, και με τη χρήση 5 και όχι 6-7 δικαστών. Δηλαδή ε, πάντοτε ε, εκδικάζονται υποθέσεις με ολομέλεια των πενταμελών. Ε, η εκλογή αντιπροέδρων επίσης επιτρέπει τη ρύθμιση του θέματος απουσίας ενός δικαστή γιατί η αντιπρόεδρη, ένας αντιπρόεδρος κάθε φορά προστίθεται όταν χρειάζεται. Οι πρώτες εμπειρίες με τα πέντε πενταμελή τμήματα είναι ενθαρρυντικές δίνει, δείχνει ότι αυξάνεται η αποτελεσματικότητα και η ταχύτητα. Το δικαστήριο λοιπόν ευνομνεί την νομοθετική, το νομοθετικό σκέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση που δέχτηκε τι προτάσει μα. Τώρα, περνάμε στο τμήμα το οποίο ακόμα δεν έχει οθετηθεί, που είναι και το πιο ακαθόδε αυτής τη μεταρρύθμισης. Δηλαδή, η πρόταση αύξηση των αριθμών, του αριθμού των δικαστών. Η κατάσταση είναι πιο δύσκολη και δημιουργεί σημαντικέ ανησυχίε. Θυμόμαστε ότι μετά από εσωτερική, πολλές εσωτερικές συζητήσεις τόσο στο Κοινοβούλιο, ε, στο, τόσο στο δικαστήριο ε, ε, όσο και στα τμήματά του, ε, είχαμε καταλήξει να επιλέξουμε από τις δύο δυνατός μας δίνει συνθήκη αυτήν της αύξησης του αριθμού των δικαστών. Το πρόβλημα δεν αφορά ε, τα σήματα τόσο πολύ ή την πνευματική ιδιοκτησία. Ε, το πρόβλημα υφίσταται στις ε, υποθέσεις που αφορούν τον ανταγωνισμό και την αύξηση του αριθμού των υποθέσεων που φτάνουν σε μας. Αν θέλουμε να έχουμε μια μόνιμη και ευέλικτη λύση, η αύξηση του αριθμού των δικαστών είναι η πιο σωστή λύση. Πολύ δε περισσότερο που με κάποια εξειδίκευση και με μέτρα, πρόσθετα μέτρα βελτίωσης της αποτελεσματικότητας, για παράδειγμα ε, ένα σύστημα για το σεβασμό των εσωτερικών προθεσμιών, θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε πάρα πολύ την αποτελεσματικότητά μας. Η πρόταση του δικαστηρίου να περάσουμε από 7 στα 39 ε, μέλη του ε, δικαστηρίου δημοσίας ε, του Γενικού Δικαστηρίου αντιστοιχεί στις πραγματικές ανάγκες. Όμως, η συμφωνία δεν έχει επιτευχθεί στο θέμα του πώς θα εκλέγονται οι δικαστές αυτοί. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να καποια κάποια κράτη-μέλη προτείνουν ένα σύστημα ε, ίδιο με, παρόμοιο με αυτό της, του Διοσμού των γενικών εισαγγελέων, άλλοι, ε, ένα σύστημα άλλα ένα σύστημα κυκλικής αναλλαγής. Ε, διάφοροι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπάθησαν αλλά δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν πολιτική συμφωνία. όμως και μάλλον η δική μας ε, αρχική πρωτοβουλία 2011 φαίνεται, φαίνεται λέω, να έχει καταπέσει, όμως δεν είναι αλήθεια. Αντιθέτως, η μεταρρύθμιση ε, του Γενικού Δικαστηρίου παραμένει ε, και δεν έχει, οι προτάσεις μας δεν έχουν χάσει την επικαιρότητά τους. Τα στοιχεία το δίνουν, δείχνουν. Βέβαια, ε, έχει μειωθεί ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων 2012 κατά 5%, αλλά αυτά τα νούμερα είναι το 2003 και πάλι αυξημένα. Ο αριθμό των εκκρεμών υποθέσεων του στις 31 Μαρτίου 2013, το τέλος δηλαδή του πρώτου τριμήνου, φτάνουν περίπου στο επίπεδο του 2010-2011. Σας υπενθυμίζω ότι αυτό ακριβώς το επίπεδο υποχρέωσε το δικαστήριο το 2011 να ζητήσει αύξηση του αριθμού των ε, δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου για να λειτουργεί αυτό ε, αποτελεσματικά το πρώτο τρίμηνο του 2013 άλλωστε ο αριθμός των νέων υποθέσεων ε, του Γενικού Δικαστηρίου ξεπερνούσε κατά 20% τον αριθμό των υποθέσεων που, είχαν, που εκδικάστηκαν την ίδια περίοδο. Ε, χαίρομαι που η, η Επιτροπή σας δίνει σημασία σε αυτό το θέμα και πήρε την πρωτοβουλία να συζητηθεί, ένα, ε, να συζητηθεί το ε, θέμα του διορισμού προς των δικαστών ανεξαρτήτως των ε, προτάσεων που είχαν στο παρελθόν. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν υπέβαλε νομοθετική πρόταση το έκανε χωρίς να υποβάλει προτάσεις ό,τι αφορά τον τρόπο διορισμού των, προς των δικαστών. Αυτό εξηγείται από το εξής. Το ε, μας δεν προβλέπει την αρμοδιότητα ε, του υποβολής τέτοιων προτάσεων. Τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα πολιτικές συζητήσεις όμως απέδειξαν ότι το θέμα της εθνικότητας των ε, δικαστών ε, έχει λάβει διαστάσεις υπερβολικές. Χωρίς ε, να θέλω να αρνηθώ τον ρόλο που παίζει η προέλευση των υποψηφίων, πιστεύω ότι αυτή δεν θα πρέπει να αποτελέσει αποφασιστική σημασία κριτήριο για το διορισμό πολύ τα περισσότερο που από την δημιουργία του το δικαστήριο ε, όλα τα κράτη-μέλη, όλες οι εθνικότητες και όλα τα ε, δικαστικά σώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκπροσωπούνται ε, αποτελεσματικά στη σύνθεση του δικαστήριου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 90% των υποθέσεων άλλωστε εκδικάζονται από τριμελή τμήματα Οπότε το να θεωρείται η εθνικότητα, η υπηκότητα ε, βασικό κριτήριο για την σύνθεση, για την, το διορισμό δικαστών, πιστεύω ότι θα δημιουργούσε εμπόδια στη λειτουργία μας. Αυτό με οδηγεί στο τελευταίο τμήμα της ε, παρουσίασής μου. Θα σας εκφράσω κάποιες ε, γενικότερες σκέψεις για το θέμα της, του διορισμού προς των δικαστών. Από πλευράς του δικαστηρίου, τρία είναι τα σημαντικά στοιχεία. Πρώτον, οι ικανότητες ε, η σταθερότητα και η ε, γεωγραφική κατανομή. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τι ικανότητε, τα προσόντα, θα πρέπει να έχουν εξαιρετικά καλή γνώση του ευρωπαϊκού δικαίου, ε, να μπορούν να μιλούν περισσότερε τη μια γλώσσα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχουν ικανότητε οργάνωση, οργανωτικέ ικανότητε. Αν λοιπόν το δικαστήριο μπορούσε να προτείνει ένα σύστημα διορισμού, θα πρότεινε περισσότερο ένα σύστημα που θα βασίζεται ε, κυρίω ένα σύστημα κυρίως αξιοκρατικό. Ε, για να μετρηθεί η ικανότητα των δικαστών, η συνθήκη της Λισαβόνας ε, έχει συστήσει την επιτροπή του άρθρου 265 ε, που θα μας επέτρεπε να κάνουμε τέτοιες επιλογές. Μετά, η σταθερότητα. Σταθερότητα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για μας. Το να μην ανανεωθεί ε, ένας ε, δικαστής για πολιτικούς και μονολόγους ε, εμποδίζει την αποτελεσματικότητα των ασιών μας. Είναι, πολύ γνω... είναι γνωστό ότι οι δικαστές που μόλις διορίζονται χρειάζονται κάποιο χρόνο για να γίνουν πλήρως λειτουργικοί και οι απερχόμενοι δικαστές είναι λιγότερο αποτελε... παραγωγικοί τους τελευταίους μήνες της θητείας τους. Να σας υπενθυμίσω ότι δεν αποκλείεται το 2013 6 ως 9 νέοι δικαστές να φτάσουν στο δικαστήριο επί ενός συνολικού αριθμού 27 δικαστών. Όμως αν ο νομοθέτης επιλέξει ένα σύστημα διορισμού των προς των δικαστών που θα εξαιρούσε καταρχήν οποιαδήποτε ανανέωση της θητείας ε, δικαστή, ε, αυτό το πρόβλημα θα οξυνόταν στα επόμενα χρόνια. Τέλος, ε, ένα ε, μια κάποια γεωγραφική ισορροπία. Σας υπενθυμίζω ότι οι διατάξεις που ε, διέπουν αυτή τη στιγμή την επιλογή προβλέπουν το δικαστήριο να, να ε, έχει μια σύνθεση γεωγραφικά ισορροπημένη που να αντικατοπτρίζει και τα νομικά συστήματα των χωρών και τον πληθυσμό των χωρών. Με άλλα λόγια, ε, θα πρέπει τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που, που προκύπτουν από την ανάγκη προσαρμογής ε, το, της ε, δομής των οργάνων στις ε, ανάγκες πραγματικότητας. Και να προβλεφθούν όσο είναι δυνατόν και οι μελλοντικές ανάγκες. Η συνθήκη της Λισαβόνας αύξησε για μία ακόμα φορά τον αριθμό των ε, θεμάτων αρμοδιότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αν ε, λάβουμε υπόψη και την εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων στις ήδη υπάρχουσες αρμοδιότητες, είναι προφανές ότι ε, το πρόβλημα θα οξυνθεί στο μέλλον και το, και το φόρτος εργασίας επίσης. Είναι λοιπόν απαραίτητο οι, οι δικαστικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να οργανωθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο εξασφαλίζοντας ότι οι δικαστικές αποφάσεις ε, θα καλύπτονται από ε, ε, νομική ασφάλεια. Ένα μοντέλο διορισμού προς τον δικαστών όπως αυτό που προτείνει η συγκεκριά σας η κυρία Τάιν μου, φαίνεται, ότι ανταποκρίνεται στις ε, απαιτήσει για ε, τι οποίες σας μίλησα και μάλιστα νομίζω ότι θα μπορούσε ε, να λύσει και ορισμένα πολιτικά προβλήματα τα οποία λαμβάνονται υπόψη. Για παράδειγμα, η λήψη, το να, υπόψη, να ληφθούν υπόψη τα θεμητά συμφέροντα των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σαφέστατη εισήγησή σας και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην εισηγήτα κυρία Αλεξάνδρα Τάιν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω θερμά τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα σχόλια του και για την συμμετοχή του και τη διευκόλυνση των διαβουλεύσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτό το η εδώ σήμερα αποτελεί μια μαρτυρία της στενής συνεργασίας και της σημασίας της ανταλλαγής απόψεων. Σήμερα θα αναφερθώ ακόμα στα εκρεμή ζητήματα της μεταρρυθμίσεως. Είναι γνωστό ότι ε, στο πρωτοβάσιμο επίπεδο το Ευρωπαϊκό Δικαστηρίο επιβαρύνεται ιδιαίτερα όχι μόνο με την εργασία βεβαίως, την αντίστοιχη εργασία των εθνικών δικαστηρίων, ανάλογη εργασία, αλλά και με τη συνθήκη της Λισαβόνας η οποία έδωσε διευρυμένες ε, αρμοδιότητες και μεγαλύτερο βάρος εργασίας. Επίσης ε, αυξήθηκε και η πίεση των ε, κρατών μελών και ανεξάρτητα από αυτή την πίεση, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε διάφορες μεταρρυθμίσεις τα τελευταία χρόνια, οι οποίε μεταρρυθμίσεις ήταν καρποφόρες. Ιδιαίτερα όταν κανείς εξετάσει τα στατιστικά στοιχεία του περασμένου έτους. Πιστεύω όμως ότι οι εσωτερικές μεταρρυθμίσεις τώρα έχουν κορεστεί. Δηλαδή, ε, υπάρχει τέτοιος φόρτος εργασίας που δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπιστεί το έργο αυτό σωστά παρά μόνο με πρόσθετους δικαστές με την προσθήκη ε, άλλων δικαστικών θέσεων. Έχω παρακολουθήσει τις εργασίες και έχω προτείνει και εγώ 12 επιπλέον θέσεις. Όσοι γνωρίζουν καλύτερα την έκθεσή μου, ε, τα, η, αριθμητική διάσταση κυμαίνεται μεταξύ 6, 9 ή 12 πρόσθετων δικαστικών θέσεων. Θα δούμε, αλλά αυτή τη στιγμή με την τρέχουσα κατάσταση το θέμα αυτό μπορεί να μείνει ανοιχτό. Το αριθμητικό δηλαδή στοιχείο, αλλά αυτό που θέλουμε εμείς να συμφωνήσουμε είναι να ε, συμφωνήσουμε όλοι να υπάρχει ομοφωνία για την αύξηση των θέσεων. Τώρα το θέμα είναι από ποια κράτη θα προέρχονται ή πρόσθετη δικαστή. Εγώ προσωπικά όταν ανέλαβα αυτό το ντοσιέ δεν είχα κατά ότι το θέμα του μεγέθους ε, του κράτους, αν είναι μικρό, μεσαίο, μικρομεσαίο ή μεγάλο, έχει τόση σημασία για την επιλεξιμότητα. Όμως ε, για τα κράτη τα ίδια είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Ε, έχουν προταθεί διάφορες κυκλικές λύσεις κυκλικών εναλλαγών. Αυτό που έχει σημασία είναι να διερωτηθούμε και να εξετάσουμε μια κυκλική διαδικασία εναλλαγή συνάδει με τις συνθήκες. Διότι σύμφωνα με τις συνθήκες μπορεί ένας δικαστής να επιλεγεί να προταθεί επανειλημμένα από ένα κράτος μέλος. Το θέμα είναι θα συμφωνήσουμε πολιτικά τα αρμόδια θεσμικά όργανα για την κυκλική εναλλαγή θα πρέπει ένας δικαστής, παραδείγματος χάρη, να εγκαταλείψει φακέλους ή υποθέσεις, διότι θα πρέπει να δώσει τη θέση του σε έναν άλλο συνάδελφο. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε και αυτή την περίπτωση, ότι ένας δικαστής που θέλει να συνεχίσει την εργασία του, να μην ονομαστεί ως επιλέξιμος από, το κράτος του ε, ε, για μια... τη θητεία του για άλλη μια φορά και εν συνεχεία να παραβιαστούν άρθρα της συνθήκης. Αυτή τη στιγμή τρέχουν, είναι σε εξέλιξη συζητήσει μεταξύ των κρατών μελών. Και το θέμα της επιλογής βάσει των κριτηρίων, των ικανοτήτων Ε, αυτά, αυτά ισχύουν για τις πρόσθετες θέσεις. Θα υπάρχει η εγγύηση της γεωγραφικής ισορροπίας, διότι βάσει της συνθήκης πρέπει να υπάρχει ένα δικαστής από, ένα, από κάθε κράτος μέλος. Το θέμα είναι τώρα ποια κράτη-μέλη, η ουσία δηλαδή του ζητήματος είναι ποια κράτη-μέλη θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής δεύτερης θέσεως. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από τις άλλες ομάδες ε, που ακολούθησαν το σκεπτικό μου και πιστεύω ότι ε, σύμφωνα με το άρθρο 255 η επιλογή των δικαστών δείχνει ότι οι δικαστές ας το πούμε έτσι δεν κρίνονται όσον αφορά τις ικανότητές τους με αυτά τα οποία μπορούν να κάνουν με τις δυνητικές τους ικανότητες αλλά αυτή η επιλογή, διαδικασία επιλογής μπορεί να κρίνει πολλούς υποψήφιους βάσει των εξαιρετικών τους ικανοτήτων. Δεν θέλουμε δηλαδή μόνο σωστά εκπαιδευμένους και καλούς δικαστές. Θέλουμε τους πιο ικανούς, τους βέλτιστους όσον αφορά τις ικανότητες εξάσκησης της εργασίας τους οι δικαστές πολλές φορές μπορούν ήδη να ε, προτείνουν την υποψηφιότητά τους. Και ο πρόεδρος του δικαστηρίου, όπως ανέφερε τώρα στην ομιλία του, ε, δεν υπάρχει εγγύηση της συνέχειας ε, και της ασφάλειας. Πρέπει να ξέρουν οι δικαστές ακριβώς πότε αρχίζει, πότε λίγη η θητεία τους, για να υπάρχει ακριβώς αυτή η νομική ασφάλεια και θα πρέπει εγκαίρως μέσα από τη διαδικασία αυτή να ανακοινώνεται το όνομα ενός νέου του αντικαταστάτη ενό νέου δικαστή. Δεν είναι δυνατόν όλα αυτά να γίνονται τελευταία στιγμή και να μην είναι γνωστά. Ε, ο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ή το, δικασ... το Πρωτοβάσμιο Δικαστήριο πολλές φορές εργάζεται με ακάλυπτες θέσεις δικαστών. Αυτό δεν είναι δυνατόν, δεν είναι επιτρεπτό. Και πολλές φορές νέοι δικαστές ναι, οι δικαστέ ε, δεν γνωρίζουν, οι οποίοι διορίζονται έτσι εντάχει α πούμε, δεν γνωρίζουν τι υποθέσει δεν είναι ενημερωμένοι. Ούτε νομίζω ότι είναι σωστό αυτό όσον αφορά την ε, νομική διαδικασία η οποία απαιτεί την ε, διευθέτηση και την εξέταση των υποθέσεων με κάποια σειρά, με κάποια τάξη. Ε, γι' αυτό λοιπόν ε, θα πρέπει και οι ίδιοι οι δικαστές να κάνουν μια αυτο, αυτοσκόπηση. Δεν μπορώ εγώ να προβλέψω ούτε να επιβάλλω κυρώσεις ε, αλίμονο, αλλά ε, θα πρέπει ένας δικαστής ο οποίος έχει τη θέση, κατέχει τη θέση του και θέλει να συνεχίσει να θέσει την υποψηφιότητά του ο ίδιος για επανάληψη της θητής και να πιέσει το κράτος μέλος του και να εξηγήσει τους λόγους τους οποίους θέλει να παραμείνει. Επίσης, μία διαδικασία δημοσίου διαγωνισμού στα κράτη-μέλη ε, είναι και αυτό ένα ε, ενδεχόμενο δεδομένου ότι καλύπτεται από τη συνθήκη και μπορεί να και νομιμοποιεί ακριβώς τον τρόπο επιλογής και διορισμού. Υπάρχουν και κράτη, μια δημόσια προκήρυξη δηλαδή των θέσεων. Υπάρχουν και κράτη όπου ο αρμόδιος υπουργό, ο υπουργό δικαιοσύνης παραδείγματος χάρη, θέλει να προτείνει ορισμένους νομικούς οι οποίοι ενδέχεται να μην είναι οι πλέον ικανοί η καλύτερη Γι' αυτό εμένω ότι θα πρέπει να γίνει δημόσια προκήρυξη της θέσης ε, σε όλα τα κράτη. Η γεωγραφική κατανομή ε, ισχύει και υπάρχει εγγύηση, δεδομένου ότι κάθε κράτος μέλος θα έχει έναν δικαστή. Ούτε υπάρχει ο κίνδυνος ότι ένα κράτος μέλος κάποια στιγμή θα έχει στο πρωτοβάσινο δικαστήριο τρεις δικαστές, διότι όπως είδαμε ε, στο για, τις, ε, για τους δικαστές που ασχολούνται με υποθέσεις ε, ε, δημοσίου δικαίου, του δημοσίου δηλαδή, των κρατών μελών, υπήρχαν δύο δικαστές οι οποίοι ήταν αρμόδιοι και έγινε μια, ένα μπλέξιμο, υπήρχε μια επικάλυψη δηλαδή και το θέμα ρυθμίστηκε και έτσι δεν υπάρχει περίπτωση να είναι τρεις δικαστές με την ίδια επικότητα Ε, στο δικαστήριο. Ε, πρέπει όλοι να φροντίσουμε και να εξετάσουμε μεγάλη προσοχή αυτές οι πρόσθετες θέσεις να ε, έχουν, να αναφέρουν υποψήφιους οι οποίες έχουν τις βέλτιστες και μέγιστες ικανότητες για να ασκήσουν τα καθήκοντά τους. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ για την, την Αλεξάνδρα Τέιν για τα, που μας μίλησε για τα κριτήρια επιλογής και θέλω να δώσω το λόγο στην Μόρα Μαγκάουαν η οποία είναι πρόεδρος του, ε, του und Συλλόγου της Αγγλίας και της Ουαλίας. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχω την ευκαιρία στο όνομα του Δικηγορικού Συλλόγου της Αγγλίας και της Ουαλίας να αναφερθώ σε ένα τόσο σημαντικό θέμα. Πώς μπορεί να συμβάλλει το, το πώς μπορούν να συμβάλλουν οι δικηγόροι ε, στην αναθεώρηση του δικαστηρίου. Επικροτούμε τον ε, νέο οργανισμό του δικαστηρίου, επικροτούμε ε, τον εξορθολογισμό που γίνεται. Για παράδειγμα, το σύστημα e-Curia για την αρχιοθέτηση είναι πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους επαγγελματίε που εργάζονται στο δικαστήριο. Χαιρόμαστε που βλέπουμε μείωση του χρόνου για τις ε, παραπομπές που τώρα πέφτει κάτω από 18 μήνες. Ε, ποιες ε, όμως είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, όπως ήδη υπόθηκε, η επαγγελματική εμπειρία των δικαστών που αποστέλλεται από τα κράτη-μέλη είναι πάρα πολύ σημαντική. Ε, πόσο μάλλον ε, τώρα που διευρύνεται το ε, ευρωπαϊκό δίκαιο και καλύπτει τομεί όπως είναι το άσυλο, το ποινικό δίκαιο και το οικογενειακό δίκαιο πολλοί σκέφτονται αποκλειστικά το ευρωπαϊκό δίκαιο ε, όταν ε, σκέφτονται ε, τους νέους διορισμούς. Θα πρέπει να είναι διαφανής η διαδικασία και αξιοκρατική. Θα πρέπει να αναζητείτε δηλαδή ο καλύτερος υποψήφιος. Θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι υπήκος μια συγκεκριμένη χώρας, μια πιο ευρεία προσέγγιση. Σίγουρα θα βοηθούσε καλύτερα πήρε στην απόδοση της δικαιοσύνης. Ε, εμείς ε, στηρίζουμε γενικά τις τελευταίες παρατηρήσεις ε, του εισηγητή. επικροτούμε τα νέα μέτρα, αλλά θα πρέπει οι δικαστές να επιλέγονται αξιοκρατικά. Θα προτείναμε τη δυνατότητα τρία κράτη-μέλη να υποβάλουν το καθένα υποψήφιο για κάθε συμπληρωματική θέση και κατόπιν η Επιτροπή του άρθρου 255 να εξετάζει τους ε, δικαστές αυτούς ε, και να τους τοποθετεί ανάλογα με τα ε, προσόντα τους. Επίσης, όσον αφορά το θέμα της κατάρτισης των δικαστών, να είμαστε ρεαλιστές. Αυτοί που διορίζονται στο Λουξεμβούργιο σπάνια θα έχουν όλες τις δεξιότητε που απαιτούνται. Μία δοκιμασμένη μέθοδος είναι να δίδεται επίσημη κατάρτιση ώστε να συνεχίζεται η επαγγελματική, ε, τους, επαγγελματική τους εξέλιξη, συγγνώμη, ώστε να ε, διευρύνονται οι δεξιότητες του και να καλύπτουν ε, νέους τομείς όπως για παράδειγμα είναι το ποινικό δίκαιο, το ασύλο ή το οικογενειακό δίκαιο. Ε, προγράμματα εκπαίδευσης ε, των δικαστών ε, με, δικαστές από άλλα κράτη-μέλη όταν φτάνουν στο δικαστήριο. Ένα σύστημα ελέγχου των νέων δικαστών από παλαιούς δικαστές. Η χρήση βέλτιστων πρακτικών από διάφορα δικαστήρια και με διαφορετική πολιετή πείρα. Το δικαστήριο θα θα πρέπει να επικεντρώνεται στην ε, παροχή πρακτικών ερμηνιών για τα εθνικά δικαστήρια. Και τα εθνικά αυτά δικαστήρια χρειάζονται καθοδήγηση για το μέλλον. Τα τα δικαστήρια θα πρέπει να χρησιμοποιούν, ε, όταν ενδείχνεται, του ε, νέου διαδικαστικού κανόνε, δηλαδή να μην έχουν ε, ακροματική διαδικασία σε κάθε περίπτωση, να μην έχουν γραπτή γνωμοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα, αλλά να δίδεται προτεραιότητα στην ποιότητα τη δικαστική απόφαση. Μπορεί να υπάρχουν περιπτώσει όπου η προφορική ακρόαση είναι πιο χρήσιμη, να χρησιμοποιηθεί δηλαδή η διαδικασία αυτή ω πρώτο το στάδιο των της εξέτασης του δικαστηρίου μιας υπόθεσης. Ε, το Γενικό Δικαστήριο μπορεί να, να χρειάζεται ε, έναν ή περισσότερους δικαστές εκ περιτροπής ε, ως διαδικαστικούς δικαστές που θα εξετάζουν όλα τα θέματα του δικαστηρίου. Μπορούν να ελέγχουν τον κατάλογο, να διανέμουν τα θέματα στο, στα διάφορα τμήματα και να εξετάζουν όλα τα διαδικαστικά θέματα. Ξέρουμε ότι το Γενικό Δικαστήριο εξετάζει την αναθεώρηση του ε, οργανισμού του, αλλά κάποια ε, θέματα θα πρέπει να επανεξεταστούν και μάλιστα πιο προσεκτικά, όπως είναι ε, το να υπάρχει κλειστή διαδικασία σε περίπτωση που κάποιος δεν γνωρίζει τα τεκμήρια της υπόθεσης. Θα πρέπει να γίνεται ανοιχτή συζήτηση όχι μόνο εντός του δικαστηρίου αλλά σε πολύ πιο ευρύ πεδίο. Οι δικηγόροι βρισκόμαστε εδώ για να βοηθήσουμε να αντιμετωπίσετε τι ε, προκλήσει αυτέ. Είμαστε οι άνθρωποι που εργαζόμαστε καθημερινά με τα θέματα αυτά. Ε, βλέπουμε, τις, ε, βλέπουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στην καθημερινή δουλειά και μπορούμε να βοηθήσουμε. Πιστεύουμε ότι υπάρχει ρόλο για του δικηγόρου σε οποιαδήποτε μεταρρύθμιση του δικαστηρίου. Η ίδρυση ΣΥΣΜΠΗ έχει εκδώσει κατευθυντήριε γραμμέ για τους δικηγόρους στο δικαστήριο σε περι περιπτώσεις ε, Προδικαστική παραπομπή, ε, αλλά πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερο να υπάρχει περισσότερη διάδραση ανάμεσα ε, στο δικαστήριο και τους δικηγόρου. Θα θέλαμε οι δικαστές να ακούν τις ανησυχίες, της επιφυλάξεις των δικηγόρων γίνονται κάποιε συναντήσει με το δικαστήριο, αλλά η επόμενη θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο. Θα πρέπει να γίνονται πιο συχνά αυτέ οι συναντήσει, ε, να είναι πιο ευρείε και να εξετάζουν περισσότερο ει βάθο τα θέματα αυτά. Μέσω πρόθεσμα η λογική απαιτεί να έχουμε μια επιτροπή περί κανόνων όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ε, οι δικαστές, ε, τα κράτη-μέλη, ε, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι δικηγόροι, να μπορούν ανοιχτά να εξετάζουν την λειτουργία του δικαστηρίου και να υποβάλουν προτάσεις για τη βελτίωσή του. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το άρθρο 253 παράγραφος 6, ο κανονισμός του δικαστηρίου απαιτεί μόνο έγκριση του Συμβουλίου των κρατών μελών δηλαδή. Κοιτώντας λοιπόν το μέλλον, τι προτείνουμε. Καταρχήν, να επιλέγονται οι καλύτεροι υποψήφοι και αυτοί να καταρτίζονται ώστε να μπορούν περαιτέρω να βελτιώνουν ε, τις δεξιότητές τους. Θα πρέπει να υπάρχει καλή ισορροπία ανάμεσα στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα στην ε, δουλειά και των δύο δικαστηρίων και το δικαστήριο θα πρέπει να στοχεύει όλοι οι ενδιαφερόμενοι που ε, συμμετέχουν στο νομικό σύστημα να συνεργαστούν ε, για ε, να βελτιωθεί η απόδοση δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ένα πρακτικό βήμα που μπορεί να γίνει είναι τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν πολιτική, να ζητούν από το, κράτος, από το δικαστήριο να διαβουλεύεται και με το Κοινοβούλιο και με τους δικηγόρους. Όπως σας είπα και πριν, ε, εμείς οι δικηγόροι βλέπουμε την ε, καθημερινή εικόνα και μπορούμε να συμβάλλουμε σε ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα για την απόδοση δικαιοσύνης. Αυτά είναι απαραίτητα ώστε ο κόσμος ε, να έχει εμπιστοσύνη στο σύστημα. Αν ο κόσμος δεν έχει εμπιστοσύνη στο σύστημα, το σύστημα δεν θα λειτουργεί σωστά. Ο Τόμ Μπίγαμ στο βιβλίο του για το κράτος δικαίου γράφει ότι μία από τις αδυναμίες του δικαστηρίου στο Λουξεμβούργο είναι η καθυστέρηση ε, η πτυχή αυτή έχει βελτιωθεί σημαντικά, αλλά ένα από τα πράγματα που ε, συνέβαλαν στις καθυστερήσεις αυτές ήταν η επιτυχία του δικαστηρίου και ο αυξανόμενος όγκος ε, καθηκόντων. Οι δικηγόροι μπορούν και είναι διατεθειμένοι να παίξουν ενεργό ρόλο στη διαχείριση των θεμάτων αυτών. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικός ο ρόλος μας για την επιτυχία του δικαστηρίου και θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στη μελλοντική επιτυχία του δικαστηρίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα θα συνεχίσουμε με ερωτήσεις των μελών μας. Ο κ. Μέσερ Σμιτ καταρχάς. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις. Από ό,τι βλέπω από το πρόγραμμα, ο κ. δεν θα είναι μαζί μας στο δεύτερο τμήμα της ε, παρουσίασης της ε, ακρόασης, οπότε δεν θα μπορέσει να πάρει μέρος στην συζήτηση. Γι' αυτό θα ήθελα να θέσω ε, ένα ερώτημα ήδη ε, για ένα τμήμα της έκθεσης, το οποίο δεν συζητήθηκε, το θέμα της διαφάνειας. Κύριε Μέσσερ θα σας παρακαλούσα, λέει πρόεδρος, να την θέσετε όταν συζητούμε το αντίστοιχο περιεχόμενο, το αντίστοιχο θέμα. Έχουμε να συζητήσουμε και τα αποτελέσματα της μελέτης. Το θέμα θα παραμείνει. Ο κύριος Μέσσεσμιτ Σίγουρα, σίγουρα θα μπορέσω να το θέσω. Η πρόεδρος. Ναι, ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Όταν έρθει η στιγμή θα σας δώσω το λόγο για να θέσετε αυτό το ζήτημα. Σε πιο κατάλληλη στιγμή. Ο κύριος Μασίτ ή ο κύριος Νταφ θέλει να μιλήσει διαδικαστικό. Κύριε Νταφ, ο κύριος Μασίπ και μετά στον κύριο Ντάφ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η παρουσίαση του Προέδρου ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Και βέβαια και η έκθεση και ο, ο ενθουσιασμός της συναδέλφου κυρία Στέιν. Την στηρίζω ανεξάρτητα από τις ε, λεπτομέρειες την υποστηρίζω γιατί ε, προσπαθεί ειλικρινά να βοηθήσει να μεταρρυθμίσει το κοινοβούλιο με την αύξηση του αριθμού, το δικαστήριο με αύξηση του αριθμού των δικαστών κλπ. Πολλές φορές ε, δεν αντιλαμβανόμαστε την πρωταρχική σημασία του δικαστηρίου στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό θα ήταν πραγματικά μεγάλο λάθος αν συνεχιζόταν. Η παρέμβαση της ε, συναδέλφου μου, λέω συναδέλφου γιατί και εγώ είμαι παλιός δικηγόρος, που εκπροσωπεί του δικηγορικού συλλόγου του Ηνωμένου Βασιλείου, ε, ήταν επίσης πολύ ενδιαφέρουσα ιδιαίτερα σε δύο θέματα. Συμφωνώ μαζί της. Ε, το υποχρεωτικό τμήμα, το, η υποχρεωτική φάση θα μπορούσε να μεταρρυθμιστεί. Ε, και ε, θα μπορούσαν, ε, θα υπάρχουν τμήματα της φάσης αυτής που θα μπορούσαν να καταργηθούν. Όμως το πιο σημαντικό είναι οι προθεσμίες. Οι προθεσμίες συνδέονται πάρα πολύ με την μετάφραση. Η μετάφραση καθυστερεί πάρα πολύ. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ενοποιήσουμε τα κριτήρια έτσι ώστε να μειωθεί το πρόβλημα της μετάφρασης διότι αλλιώς είναι προφανές ότι ε, η μετάφραση έχει σχέση με τα δικαιώματα της υπεράσπισης. Ε, αλλά το δικαστήριο είναι ε, βασικό όργανο και όπως λέει και η Αλεξάνδρα Τέιν, θα πρέπει ε, οτιδήποτε γίνεται, οποιασδήποτε διαδικασίες να είναι πριν οτιδήποτε κάνουμε μάλλον, οτιδήποτε νομοθετήσουμε θα πρέπει να γίνεται πριν την εκδίκαση ε, και πριν παρουσιαστούν τα προβλήματα. Ο Λόπεθ Ιστούρη δεν είναι παρόν σήμερα, αλλά ε, έχει πει επανειλημμένως κάτι πολύ σημαντικό, ότι η ποιότητα ε, θα πρέπει να εξασφαλίζεται από την αξιοκρατία. Ε, το είπε και η Αλεξάνδρα Τέιν ότι Υπάρχουν κριτήρια όπως η γεωγραφική ισορροπία, αλλά τελικά στο κοκτέιλ αυτό, στο τελικό αποτέλεσμα της, του διορισμού, του ορισμού των δικαστών, ε, οι ορισμοί ε, δεν θα πρέπει ε, η αξιοκρατία να πληγεί. Θα ανεξαρτήτως της προέλευσης των δικαστών θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ποιότητά τους. Τέλος, Α, έγινε και μια αναφορά στην... Ε, ε, στην ε, διαδραστικότητα. Και μεταξύ δικηγόρων και δικαστών. Είναι πράγματι σημαντικό να υπάρχει και να είναι αποτελεσματική. Ε, διότι οι μερικοί δικηγόροι σε ορισμένε χώρε ε, δεν έχουν αυτή την παράδοση και ε, ενδεχομένως ε, δεν ακολούθησαν αυτή την οδό στο παρελθόν. Τέλο να πω το εξή. Η πρώτη φράση του Προέδρου ήταν ότι θα χρησιμοποιήσει τα γαλλικά ως γλώσσα του δικαστηρίου. Πράγματι, στην επίσκεψη που κάναμε στην προηγούμενη θητεία ε, αντιληφθήκαμε ότι ε, η, η, αντιληφθήκαμε τη μεγάλη σημασία της κοινή γλώσσας, της μιας κοινή γλώσσας για να για να ε, αποφευθεί η παρουσία ε, διερμηνέων ε, κατά τη διάρκεια των διασκέψεων. Θυμάμαι ότι ένας ε, δικαστής που νομίζω ήταν Κύπριος που έφτασε στο δικαστήριο χωρίς να ξέρει γαλλικά έκανε μια τιτάνια προσπάθεια ε, να μάθει γαλλικά και τελικά ε, οι αποφάσεις του και το σκεπτικό τους είναι εξαιρετικό στα γαλλικά πια. Το θέμα είναι το εξής η, γλώσσα θα πρέπει να αποτελέσει κριτήριο για την επιλογή των δικαστών. Θα πρέπει δηλαδή να έχουν όχι μόνο γνώση της γαλλικής γλώσσας αλλά και βαθιά γνώση του δικαίου και της γλώσσας που χρησιμοποιείται στα δικαστήρια των γαλλόφωνων χωρών. Γιατί ο Κύπριος δικαστής τα κατάφερε, αλλά μπορούν να τα καταφέρουν όλοι. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα, μήπως θα έπρεπε όλοι οι υποψήφοι να γνωρίζουν γαλλικά γιατί αλλιώς θα αντιμετωπίσουν πολλέ δυσκολίε ή τουλάχιστον αν δεν είναι επίσημο κριτήριο να το γνωρίζουν ότι θα βρουν τέτοιε δυσκολίε μπροστά του. Σα ευχαριστώ κύριε Μασίφ. Ο κύριο Νταφ έφυγε οπότε δίνω το λόγο στον ε, συνάδελφο κύριο Τσβίφκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τη σαφέστατη εισήγησή του και για τις προσδοκίες που εξέφρασε για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε η κυρία Μαγκάου για τις αδυναμίες ε, του δικαστηρίου και των δικαστηρίων γενικά. Το μεγάλο πρόβλημα είναι οι καθυστερήσεις από την αρχή της διαχείρισης ενός φακέλου μέχρι τη στιγμή της απόφασης. Βεβαίω, ο νόμος θα πρέπει να ενεργεί γρήγορα, να έχει γρήγορο αποτέλεσμα και βεβαίω δεν θέλουμε μία μακρά διαδικασία ε, μεταξύ της αρχής μιας υποθέσεως και του τέλους. Ε, διότι εδώ ε, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που έχουν σχέση με την οικονομική ζωή, εμπορικές συναλλαγές, εμπορικές δικογραφίες με εμπορικής φύσεως και εμπορικά θέματα. Και οι εισηγόμενοι απαιτούν γρήγορες αποφάσεις. Τώρα δεν θα κρίνω εγώ ε, το, το, το, επιχείρημα ότι περισσότεροι δικαστές θα μειώσουν την καθυστέρηση που σημειώνεται στην εκδίκαση των υποθέσεων. Όμως δεν σύμφωνο με την εξής δήλωση ότι ένα κράτος μέλος θα ονομάσει ή ονομάζει ορισμένες φορές υποψήφιους χαμηλότερων ικανοτήτων. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι σωστό. Μειωμένων ικανοτήτων. Δεν είναι σωστό να το λέει κανείς αυτό, διότι αποτελεί τιμή για κάθε κράτος μέλος να ονομάζει και να έχει ως εκπρόσωπο τον καλύτερο, τον βέλτιστο. Βεβαίω μπορεί να υπάρχει κάποια ανησυχία για τα μικρότερα κράτη-μέλη όπου να υπάρχει κάποια έλλειψη ε, γλωσσικών γνώσεων ή ε, να υπάρχουν κάποιες ελλείψεις στη γνώση του ε, του υλικού ή όλων των περιπτώσεων να μην υπάρχει μια ολοκληρωμένη ας πούμε γνώση αλλά ε, μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τις μικρότερες χώρες όμως δεν μπορούμε να πούμε ή να ε, υποθέσουμε ότι είναι αναπόφευκτο ότι ορισμένοι δίκαστες θα είναι χαμηλό, ε, πιο μειωμένων ικανοτήτων ή θα είναι οι ε, αυτοί που προτιμήθηκαν από κάποιον ή κάποιους υπουργούς δικαιοσύνης ε, είναι, είναι κύρος, αποτελεί μεγάλο κύρος και μεγάλη τιμή για ένα κράτος μέλος να έχει τον εκπρόσωπό του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Οπότε ε, η επικρατεί η αξιοκρατία στην επιλογή. Υπερισχύει λοιπόν το αξιοκρατικό κριτήριο. Γι' αυτό μία γεωγραφική κατανομή των δικαστών δεν, δεν επηρεάζει την ποιότητα. Τώρα, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα με τις πρόσθετες θέσεις, διότι ο των δικαστών δεν θα αντιστοιχεί ακριβώς στον αριθμό των κρατών μελών. Και το άλλο ερώτημα είναι, μπορούμε να έχουμε την πολυτέλεια να αυξήσουμε τόσο πολύ τον αριθμό των δικαστών, την οικονομική δυνατότητα. Την έχουμε. Κύριε Πρόεδρε του Δικαστηρίου, έχω μία ερώτηση. czy dzisiaj w sprawozdaniu e, koleżanki czy w e, Υπάρχουν ορισμένοι μηχανισμοί που προτείνονται στην έκθεση της κυρίας Τάιν στη συζήτηση που γίνεται στο Συμβούλιο. Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιος προτινόμενος μηχανισμός ε, με τον οποίο δεν συμφωνείτε, ο οποίος πιστεύετε ότι δεν είναι σωστός και δεν συνάδει με τις αρχές ε, της επιλογής των βέλτιστων δικαστών, των ικανοτέρων. Μήπως νομίζετε ότι υπάρχει κάποιος μηχανισμός προτινόμενος, κάποια διάταξη, κάποια ε, ιδέα που προτείνετε την οποία θα πρέπει να αποκλείσετε. Και θα Ήθελα τώρα να ε, προτείνω να ξεπεράσουν τα κράτη-μέλη τις, τις πολιτικές πτυχές και να επιλέξουν τους ικανότερους για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να δώσω την ευκαιρία στον ε, κύριο Σκουρή να απαντήσει στις ερωτήσεις αυτές. Παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να σας πω τη γνώμη μου για διάφορα πράγματα τα οποία εκτέθηκαν. Ε, ελπίζω να μην ξεχάσω τίποτα. Το θέμα της επιλογής των δικαστών. Που επίσης αφορά το ακαθόδες πρόβλημα του αν υπάρχουν οι αναφέρονται μηχανισμοί στο, στην πρόταση, τους οποίους θεωρούμε ως ασύμβατους με το σύστημα ή ασύμβατους με τις ανάγκες ε, του δικαστηρίου. Θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι το Συμβούλιο που είναι αρμόδιο και πιο συγκεκριμένα η συνεδρίες των εκπροσώπων των κρατών μελών που ε, είναι το Συμβούλιο, λέω, ε, και πιο συγκεκριμένα η Επιτροπή των Εκπροσώπων των Κρατών Μελών που διορίζει τους ε, δικαστές. Συνεπώς το δικαστήριο δεν έχει αρμοδιότητα να λάβει, να λάβει πρωτοβουλία, να κάνει προτάσεις. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε δεν κάναμε πρόταση στο παρελθόν σε ό,τι αφορά το θέμα του ορισμού των δικαστών. Το θέμα εκφεύγει των αρμοδιοτήτων μας και δεδομένου το δικαστήριο έχει ως βασικό καθήκον να ελέγχει το κατά πόσον τα όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση σέβονται τι αρμοδιότητε, τι αντίστοιχε αρμοδιότητες, ε, είναι προφανές πως ε, θα ήταν πολύ άσχημο μήνυμα το ίδιο το δικαστήριο να μην ε, σέβεται την κατανομή αρμοδιοτήτων. Όμω, εν τω μεταξύ Πέρασαν δύο χρόνια συζητήσεων, αναπτύχθηκαν μοντέλα, το ένα μετά το άλλο. Το σύστημα κυκλικής αναλλαγής, για παράδειγμα. Παρόλες αυτές τις προσπάθειες δεν πετύχαμε. Με αυτό το φόντο θέλουμε να ενθαρρύνουμε και μέσω της σημερινής συζήτησης και γενικότερα στο πλαίσιο των συζητήσεων του Κοινοβουλίου ο, να, λέω, να προωθήσουμε μια λύση με εξαίρεση κάποιων κριτηρίων, με αποκλεισμό κάποιων κριτηρίων. Όχι να κάνουμε πλήρη πρόταση σε ό,τι αφορά τον διορισμό των των δικαστών, αλλά να αποκλείσουμε τουλάχιστον κάποια κριτήρια. Και πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να αναφερθούν ή αντιθέτως να υπογραμμίσουμε ποια θα έπρεπε να είναι τα βασικά κριτήρια. Και τα βασικά κριτήρια για μας είναι η αξιοκρατία που θα εξασφαλίσει την ποιότητα. Θα πρέπει αυτό το κριτήριο να είναι η βάση πρόταση που θα προέρχεται από τα κράτη-μέλη. Επί των υπολείπων δεν μπορώ και δεν πρέπει να κάνω πιο συγκεκριμένες προτάσεις. Πιστεύω ότι αν τα κράτη-μέλη δεχθούν ότι οι ορισμοί θα πρέπει να είναι αξιοκρατικοί και όχι επί τη βάση της ε, εθνικής προέλευσης, μπορούμε να βρούμε σύστημα, συστήματα, τα οποία θα είναι τα πιο κατάλληλα για να ε, εφαρμόσουν την πράξη αυτό τον κανόνα. Δεύτερο θέμα, το ζήτημα της γλώσσας εργασίας. Υπάρχουν υποψήφοι προφανώς που δυσκολεύονται πολύ περισσότερο με τα γαλλικά. Είναι σαφές ότι ε, ε, είναι σημαντικό οι διασκέψεις, διασκέψεις να γίνονται σε μία γλώσσα. Δεν είναι δυνατόν να διασκεπτόμεθα σε πολλές γλώσσες γιατί το αποτέλεσμα είναι διαφορετικό. Για μας είναι λοιπόν πρωταρχική σημασία ε, η ύπαρξη μια κοινή γλώσσα. Όχι, δεν έχει σημασία ποια γλώσσα, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε να διασκεπτόμεθα σε μία γλώσσα. Αυτή τη στιγμή είναι τα γαλλικά. Ε, Από την αρχή ήταν τα γαλλικά. Όμως, τώρα ποιοι είναι οι όροι, ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Αν διαβάσετε την έκθεση του, της Επιτροπής 255 που βασίζεται σε μια εμπειρία 50 περίπου υποθέσεων είναι προφανές ότι ε, δεν χρησιμοποιούν τέλεια τα γαλλικά ε, όλοι οι υποψήφοι και παρόλα αυτά ε, δεν απέτυχαν να εκλεγούν πολλοί από αυτούς στο δικαστήριο. Είναι σαφές ότι θα πρέπει κανείς να καταλαβαίνει τα γαλλικά. Αλλά δεν είναι απαραίτητο να τα μιλάει τέλεια. Και είναι σαφές αυτό. Αν κάποιος θέλει να γίνει μέλος σε ένα όργανο που η γλώσσα εργασία είναι μια συγκεκριμένη γλώσσα, γλυκά, γαλλικά, γερμανικά, θα πρέπει να κάνει μια προσπάθεια να τη μάθει. Έτσι δεν είναι. Οποιοςδήποτε νομικός, ε, καλός, μπορεί να τη μάθει τη γλώσσα. Συνεπώς, δεν χρειάζεται μια τέλεια γνώση της ε, γαλλικής. Και αυτό αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα της Επιτροπής 255. Όμως, θα πρέπει τουλάχιστον να καταλαβαίνει καλά τα γαλλικά ο υποψήφιος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ε, σχέσεις μας με τα νομικά επαγγέλματα. Ασφαλώς θα μπορούσαν να ενταθούν οι σχέσεις αυτές, να συσφιχθούν και χαιρόμαστε που η CCPA έστειλε πριν από δύο εβδομάδε μια επιστολή στο Συμβούλιο ακριβώς για το θέμα της ε, ε, ε δικαστών. Και η CCP ακριβώς έλεγε ότι το βασικό κριτήριο θα πρέπει να είναι η ποιότητα. Συμφωνούμε και χαιρόμαστε για αυτή την ε, πρωτοβουλία. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα βελτιώσει σίγουρα τη σχέση ανάμεσα στο δικαστήριο και τα νομικά επαγγέλματα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Τάιν. Ναι, πολύ σύντομα. Τα κρότη μελη τελικά κρύβονται πίσω από τα συμφέροντά τους ε, κατά την, ε, κατά την εναλλαγή των ε, δικαστών. Λένε ότι έχουν πολλούς νομικούς και γι' αυτό έχουν μεγαλύτερη ομάδα από τους οποίους μπορούν να επιλέξουν ε, λένε τα μεγάλα. Τα μικρά κράτη-μέλη έχουν λιγότερους νομικούς, ωστόσο ε, είναι ε, εξειδικευμένοι. Για παράδειγμα η Μάλτα έχει λιγότερους από 50 δικαστές έχει βέβαια καθηγητές ε, και ε, νομικών και δικηγόρους, ε, από τους οποίους θα μπορούσε να βρει κανείς σε μια κατάλληλη προσωπικότητα. Και όταν μιλάμε για τις δεξιότητες, τότε και, και τα μεγάλα κράτη-μέλη και τα μικρά κράτη-μέλη ε, μπορούν ε, να αποδείξουν ε, ότι έχουν δίκιο. Δηλαδή τα μικρά μπορούν να αποδείξουν ότι ακόμα και από περιορισμένο αριθμό μπορούν να προτείνουν κάποιον κατάλληλο άνθρωπο και τα μεγάλα κράτη-μέλη μπορούν να αποδείξουν ότι παρά το μεγάλο μέγεθος του νομικού πληθυσμού μπορούν να επιλέξουν κάποιον κατάλληλο. Το ότι ένα κράτος μέλος είναι μεγάλο ή μικρό δεν σημαίνει ότι ε, υπάρχει ποσοστό τόσων ε, καταλήλων ε, δικαστών. Και γι' αυτό η ποιότητα για μένα είναι το μόνο επιχείρημα σε αυτή την αντιδικία ανάμεσα στα μεγάλα και τα μικρά κράτη-μέλη. Και το θέμα της εναλλαγής μπορεί να απαντηθεί ακριβώς έτσι. Και επίσης ε, όσον αφορά τη γλώσσα, να πω ότι για μένα είναι σημαντικό ε, να υπάρχει μία ε, γλώσσα η οποία να είναι αρκετά σαφής για τις νομικές χρήσεις και χρησιμοποιούμε τα γαλλικά είδαμε ότι τώρα με την ε, οικονομική κρίση ε, τα αγγλικά μπορεί να τα ερμηνεύσει κανείς ε, όπως θέλει σε κάποιες περιπτώσεις. Γι' αυτό αν από την αρχή είχαμε μια πιο σαφή γλώσσα, μπορεί να είχαμε αποφύγει μερικά από τα προβλήματα της οικονομικής κρίσης. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Κόβαν. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα επαναλάβω την πρότασή μας. Εμείς ως επαγγελματίες βλέπουμε τα καθημερινά προβλήματα και μπορούμε να βοηθήσουμε σε πρακτικό και ρεαλιστικό επίπεδο. Συμφωνώ απόλυτα με τα όσα υπόθηκαν σχετικά με την ανάγκη για ποιότητα σε οποιοδήποτε δικαστή, από οποιοδήποτε κράτος μέλος ε, τοποθετείται σε οποιαδήποτε θέση ποιότητα και το να έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο για την κατάλληλη δουλειά. Αυτά θα πρέπει να είναι τα βασικά πράγματα που θα πρέπει να σκεφτούμε. Ε, βέβαια, είναι απόλυτα σωστό αυτό που μόλις υπόθηκε. Το γεγονός ότι ένα μικρό κράτος μέλος μπορεί να παρουσιάσει τελικά μόνο δύο ή τρεις ε, υποψηφίους, δεν μειώνει την ποιότητά τους, ε, μόνο τον αριθμό περιορίζει και θα πρέπει ε, να λάβουμε υπόψη την δίκαιη εκπροσώπηση όλων των κρατών μελών. Επαναλαμβάνουμε το αίτημά μας για ποιότητα που θα πρέπει να ισχύει περισσότερο από την υπηκότητα, αλλά και τα δύο θα πρέπει να ληφθούν υπόψη επαναλαμβάνουμε το αίτημά μας να συμμετέχουμε στην καθημερινή αντιμετώπιση προβλημάτων και, στην, ε, και στο μελλοντικό καθορισμό ε, κανόνων για να λυθούν τα προβλήματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στο επόμενο, στην επόμενη παρουσίαση. Ζήτω συγγνώμη. Μόλις μου είπαν ότι υπάρχει εδώ και εκπρόσωπο τη Κομισιόν, ε, στον οποίο επίσης θα ήθελα να δώσω το λόγο. Καλωσορίζω τον κύριο Κεπέν και θα ήθελα να του δώσω το λόγο διότι είμαι βέβαιη ότι και η Κομισιόν ε, μπορεί να ε, συνεισφέρει στη συζήτηση πάνω στο θέμα αυτό. Παρακαλώ. Merci, Madame la Présidente. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η Κομισιόν είναι ε, αναφαντών υπέρ της προτάσεως που συζητούμε. Χαιρόμαστε που βλέπουμε να υφίσταται σύγκληση απόψεων μεταξύ των ε, ομιλητών, μέλη του Κοινοβουλίου και πρόεδρου του Δικαστηρίου, γιατί Όλε αυτέ οι γνώμες συμπίπτουν με την άποψη τη ε, Κομισιόν σε ό,τι αφορά την αρχική πρόταση του δικαστηρίου. Αυτό θα πω μόνο. Μια γενική σκέψη δηλαδή. Υποστηρίζουμε πλήρω τι προσπάθειε σα και είμαστε στην διάθεση όλων των οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια συνένεση. Ευχαριστώ. Και έτσι προχωρούμε στο επόμενο μέρος ε, της ακρόασης τις ε, διαφορετικές ε, γνώμες. Και η... θα μας μιλήσει πρώτα η κυρία Ρόζα Ραφέλη. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω αυτή τη μελέτη η οποία έγινε από το Τμήμα Εσωτερικών Πολιτικών εσωτερικής στρατηγικής, τμήμα Γ. Πριν ε, μπω στην ουσία της μελέτης, θα πρέπει να δώσω ορισμένες εξηγήσει για τον ορισμό του separate opinion, διαφορετική γνώμη. Είναι αυτό, αυτός ο όρος σημαίνει ότι υπάρχει διαφορετικές γνώμες όσον αφορά την απόφαση, την, τελική απόφαση. Υπάρχει μία διαφωνούσα μειοψηφία και μία ε, άλλη ομάδα η οποία έχει σύμφωνη γνώμη. Λοιπόν, ε, η διαφωνούσα μειοψηφία ε, διαφωνεί με την απόφαση του δικαστηρίου και το θέμα αυτό είναι επίμαχο. Οπότε επιτρέπεται η δημοσίευση της απόφασης του δικαστηρίου σε ορισμένες χώρες, ενώ σε άλλες χώρες απαγορεύεται τελείως. Και αυτή η διαφορά μεταξύ του separate opinion και της ε, διαφωνούσας ή μειοψηφούσας ομάδας και της σύμφωνης γνώμης ισχύει σε ορισμένες χώρες και γι' αυτό θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να επιτρέψουμε τη δημοσίευση των ε, διαφορετικών ε, αποφάσεων. Υπάρχουν 7 κράτη-μέλη όπου δεν επιτρέπεται η δημοσίευση των ε, separate opinions, διότι υπάρχει μεγάλη αντίρρηση στο, επί της δημοσιεύσεως και αποτελεί ποινικό αδίκημα στην, στο Βέλγιο και στην Ιταλία μάλιστα ποινικοποιείται η δημοσίευση αυτή ως αδίκημα. Σε άλλες χώρες τα separate opinions μπορούν να δημοσιευθούν. Όχι όμως πάντα σε όλες τις περιπτώσεις. Σε 13 κράτη-μέλη, που τα μέλη που βλέπετε με πράσινο οι διαφορετικές ε, αποφάσεις δημοσιεύονται, αν και σε ποινικέ ε, περιπτώσεις, ε, σε ποινικέ υποθέσεις η δημοσίευση περιορίζεται, είναι υπό όρους. Υπάρχουν έξι κράτη-μέλη όπου τα separate opinions δημοσιεύονται μόνο όταν πρόκειται περί συνταγματικών υποθέσεων, ενώ οι συνήθεις δικαστές ή δικαστές που ασχολούνται με τα συνήθι θέματα δεν επιτρέπεται να δημοσιεύσουν τα separate opinions. Και στην Ιρλανδία τα separate opinions δημοσιεύονται μόνο στις συνήθει υποθέσεις ενώ στα συνταγματικά ή στο συνταγματικό δίκαιο δεν επιτρέπεται να δημοσιευθούν. Είναι λοιπόν σημαντικό να σας εξηγήσω ορισμένα επιχειρήματα υπέρ και κατά των separate opinion. Είναι μια θεωρητική συζήτηση του θέματος εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκοί έχουν προβάλει επιχειρήματα κατά των separate opinions. Το πρώτο επιχείρημα είναι ότι αυτού του είδους οι αποφάσεις μπορούν να υπονομεύσουν την ανεξαρτησία των δικαστών. Ιδιαίτερα την ανεξαρτησία τους ε, κατά, από εξωτερικές πιέσεις. Ιδιαίτερα στα πλαίσια της διεθνούς δικαστικής αρμοδιότητας, διότι βεβαίως οι δικαστές διορίζονται και μπορούν να επαναδιοριστούν από εθνικέ κυβερνήσεις. Και αυτό το οποίο οι εμπειρογνώμενες φοβούνται είναι ότι ένας δικαστής ο οποίος έρχεται προς το τέλος της θητείας τους μπορεί να υποκύψει ε, σε πιέσεις και να εκδώσει μια separate opinion η οποία θα συνάδει με την ε, γνώμη της εθνικής του κυβέρνησης. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβλημα. Διότι, ας πούμε, στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο επαναδιορισμός των δικαστών ε, έχει αναθεωρηθεί. Οι κανόνες έχουν αναθεωρηθεί. Διότι στόχος είναι να υπάρξει εγγύηση για την ανεξαρτησία των δικαστών ανεξαρτησία των αποφάσεων των δικαστών. Επίσης υπάρχει ένας άλλος ε, φόβος ότι μπορεί να υπονομευθεί η απόφαση, η ουσία της απόφασης και δεν θέλει ο δικαστής να δώσει σύμφωνη γνώμη διότι είχε διαβλέψει ότι υπάρχουν διαφορετικές αναλλακτικές λύσεις για την απόφαση. Ε, το, το άλλο επιχείρημα κατά των separate opinions είναι υπονομεύουν τη σαφήνεια. Όταν οι διάδικοι πηγαίνουν στο δικαστήριο θέλουν να, βρουν μια, θέλουν να καταλήξουν σε μια σαφή απόφαση, ξεκάθαρη απόφαση. Δεν θέλουν αμφιλεγόμενες αποφάσεις που μπορεί να είναι ε, προσ, ε, προσβλητές. Και ένα ε, άλλο επίσης πρόβλημα όσον αφορά τα separate opinions είναι ότι κατά κάποιον τρόπο απειλεί τη συναδελφικότητα των δικαστών. Διότι οι δικαστές που ασχολούνται με μία υπόθεση, όταν ξέρουν ότι υπάρχει μία δυνατότητα separate opinion, μπορεί να χωριστούν στην ε, πλειοψηφία η οποία λαμβάνει, γνώμη, λαμβάνει θέση στην, και συμμετέχει στην έκδοση της απόφασης και στη μειοψηφία που δεν συμμετέχει. Και τέλος υπάρχει και η διάσταση του χρόνου και των που καταλαβαίνετε είναι σημαντικό πρόβλημα όταν έχουμε και το γλωσσικό, ε, τη γλωσσική πτυχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με όλες τις μεταφράσεις που πρέπει να γίνουν. Τώρα, υπάρχουν και επιχειρήματα υπέρ των separate opinions. Το βασικό επιχείρημα υπέρ είναι η διαφάνεια σε ε, πολλοί εμπειρογνώμονες πιστεύουν ότι θα βοηθήσει στην ε, άσκηση των ε, καθηκόντων και θα εντείνει την διαφάνεια. Επίσης θα αυξήσει τον δημοκρατικό έλεγχο για το πώς ασκείται η δικαστική εξουσία. Ορισμένοι άλλοι υπέρμαχοι πιστεύουν ότι οι separate opinions αυξάνουν το επίπεδο του διαλόγου μεταξύ των ε, δικαστηρίων και των ε, νομικών, των ε, επαγγελματιών, δικηγόρων και κλπ. Και ότι υπάρχει περίπτωση στο νόμο να αλλάξει το διδικασμένο των δικαστηρίων ή ορισμένοι δικηγόροι μπορεί να προβάλλουν επιχειρήματα ορισμένων νομοθετών και στο μέλλον να αλλάξει ακριβώς ε, η πορεία του δεδικασμένου. Άλλο ένα επιχείρημα των separate opinions είναι ότι προστατεύει αυτή η δυνατότητα την ελευθερία των δικαστών και ενισχύει την ακαιρεότητα του δικαστικού σώματος, διότι οι δικαστές δεν είναι υποχρεωμένοι ντε και Sony να συνυπογράψουν μια απόφαση. Έχουν μια άλλη επιλογή. Και επίσης ε, λένε οι υπέρμαχοι ότι μπορεί να εκδοθούν ε, σαφέστερες και καλύτερες αποφάσεις. Διότι όταν τα separate opinions ε, κυκλοφορούν και μπορούν, είναι προσβάσιμες πριν από την απόφαση, μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα της τελικής απόφασης, διότι οι δικαστές μπορεί να λάβουν υπόψη τις, ε, τους διαφωνούντες της μειοψηφίας και να ε, λάβουν υπόψη τις απόψεις τους. Και έτσι λοιπόν η απόφαση μπορεί να είναι πιο ολοκληρωμένη, πιο ισχυρή και πιο διαφανής και σαφής. Άρα θα είναι εν τέλει πιο πιστική για τους ε, διαδίκους. Τώρα, τι γίνεται στα διεθνή και υπερθνικά δικαστήρια. Υπάρχει γενικά μια τάση να επιτραπεί στους διεθνείς δικαστές να δημοσιεύσουν separate opinions. Αυτή είναι η πρακτική από το διεθνές ε, δικαστήριο και όλα τα ε, δικαστικά σώματα να επιτρέψουν αυτές τις separate opinions. Σε μερικές περιπτώσεις επιτρέπεται η δημοσίευση των αποφάσεων αυτών, παραδείγματο χάρη στο, στον ΠΟΕ και σε ορισμένα άλλους διεθνείς φορείς δεν προβλέπονται σαφώς δηλαδή τα separate opinions. Τώρα ποιος είναι ο λόγος αυτού του εξαιρετικού καθεστώτος ή επιτρέπονται κατ' Πρέπει να λάβουμε υπόψη το νομοθετικό και ε, δικαστικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό του. Εμείς αυτή τη στιγμή προτιμούμε προδικαστικές τη διαδικασία των προδικαστικών αποφάσεων. Ε, έτσι ώστε κάποιος που προσφεύγει στο δικαστήριο ή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, έχει μία ολοκληρωμένη εικόνα από, τις εθνικές, από τα εθνικά δικαστήρια προδικαστικών αποφάσεων. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λοιπόν μπορεί να εξετάσει ε, προδικαστικές εθνικές αποφάσεις και να τις ε, ενσωματώσει στο σκεπτικό. Έτσι μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι και οι εθνικοί δικαστές εμπιστεύονται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και παραπέμπω σε αυτό, αλλά είναι επίσης απαραίτητο, διότι από τη στιγμή που το δικαστήριο εκδίδει απόφαση, η απόφαση αυτή, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δηλαδή, θα, γίνει, θα είναι σεβαστή και θα εφαρμοστεί, θα υλοποιηθεί, δηλαδή θα ισχύσει στο εθνικό, στην εθνική επικράτεια. Υπάρχει βέβαια και το πρόβλημα των νομικών ε, του νομικού περιβάλλοντος. Σε ορισμένες χώρες αυτά τα separate opinions είναι τελείως άγνωστα. Και ένας εθνικός δικαστής όταν λάβει στα χέρια του μία απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που περιλαμβάνει και separate opinions μπορεί να επιφέρει σύγχυση και να μην γνωρίζει τι να κάνει. Αυτή τη στιγμή επίσης συζητείται στο ακαδημαϊκό και επαγγελματικό περιβάλλον το ρόλο του Ευρωπαϊκού Δικοστηρίου και γενικά τη δυνατότητα εισαγωγής αυτού του καθεστώτος ε, των separate opinions. Έχουν, γίνει, έχουν ακουστεί πολλά επιχειρήματα τα οποία στοχεύουν ειδικά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ορισμένοι λοιπόν εμπειρογνώμονες του τομέα έχουν επικρίνει το στυλ και τα επιχειρήματα στα οποία βασίζονται οι αποφάσεις και ορισμένες φορές οι αποφάσεις είναι αφιλεγόμενες και δυσνόητες. Κατά την άποψή τους λοιπόν αυτό το πρόβλημα μπορεί να ξεπεραστεί με την εισαγωγή των ε, διαφορετικών ε, αποφάσεων, των separate opinions. Πρέπει να βρεθεί λοιπόν στο τέλος μια κοινή απόφαση των δικαστών. Πάντως, οι εμπειρογνώμονες του κλάδου έχουν τονίσει και τη σημασία του ρόλου του Γενικού Εισαγγελέα και έχουν πει ότι το ιστορικό της δημιουργίας αυτής της θέσεως είναι να υπάρξει ένα ένας αντικαταστάτης, ένας αναπληρωτής που θα κρίνει σε περίπτωση των separate opinions. Πίσω δηλαδή από την τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου να γίνει μία συζήτηση ε, επί τη βάση των separate opinions. Τώρα όσον αφορά το στοιχείο της συναδελφικότητας, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι γνωστό ότι έχει μια πάρα πολύ συναδελφική και καλή ατμόσφαιρα και συνεργασία μεταξύ των δικαστών. Είναι θα έλεγα μια εξαιρετική περίπτωση ενός δικαστηρίου και υπάρχει ε, ο φόβος ότι με την εισαγωγή της ε, δυνατότητας separate opinions θα υπονομευτεί αυτή η συναδελφικότητα. Επίσης υπάρχει το επιχείρημα της ισχύω, της εξουσίας των δικαστών, το οποίο είναι πολύ σημαντικό στο νομοθετικό και δικαστικό, στο δικαστικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου το δικαστικό σώμα πρέπει να συνεργάζεται συνέχεια και μπορεί ενδεχομένω αυτό το νέο καθεστώς να υπονομεύσει την ανεξαρτησία και την αξιοπιστία των δικαστών. Αυτά ήταν τα υπέρ και τα κατά επιχειρήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μέσσερ Σμίτ έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Γραμματεία που μας έδωσε το σημαντικό και ενδιαφέρον αυτό υλικό εισαγωγικά να πω ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει κανένα κράτος μέλος το οποίο να μην γνωρίζει τις διάφορες γνώμες. Διότι όλα τα κράτη-μέλη συμμετέχουν στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και εκεί επί πολλά χρόνια ε, έχουμε ε, το καθεστώς της διάφωνη γνώμης. Ε, Όλοι λοιπόν ε, οι ε, επαγγελματίες, οι δικαστές ε, στα κράτη-μέλη που πρέπει να αξιοποιήσουν αυτές τις αποφάσεις του Στρασβούργου γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται. Το θέμα είναι εάν το ΔΕΚ θα πρέπει να παραμείνει το μόνο διεθνές δικαστήριο χωρίς αυτό το μέσο διαφάνειας απέναντι στους πολίτες του. Και θα ήθελα σύντομα να αναφερθώ σε κάποια επιχειρήματα που ακούσαμε. Καταρχήν, όπως αναφέρεται και στην έκθεση, υπάρχει το θέμα της ε, αυθεντίας. Νομίζω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε αν είναι δίκαιο ε, έστω και μία μικρή πλειοψηφία του σώματος των δικαστών ε, να ε, εποφελούνται από την αυθεντία του συνόλου του δικαστηρίου. Και το επιχείρημα αυτό μπορεί να πάει προς και τις δύο κατευθύνσεις. Δεν υπάρχει λόγος μικρή πλειοψηφία του σώματος των δικαστών να έχουν τελικά την απόλυτη, να χαίρουν της απόλυτης αυθεντίας. Και δεύτερον για τους ε, δικηγόρους. Ε, νομίζω ότι η έλλειψη διαφάνειας ε, στη συζήτηση των δικαστών οδηγεί σε λιγότερη συνειδητοποίηση και γι' αυτό υπάρχει δυσκολία χρήσης αυτών των διάφορων γνωμών διότι οι επαγγελματίες δεν γνωρίζουν τις, οι δικηγόροι δηλαδή δεν γνωρίζουν τις συζητήσεις που έχουν διεξαχθεί μεταξύ των δικαστών. Και το άλλο θέμα που θα πρέπει να συζητήσουμε είναι τι ακριβώς είναι η διάφωνη γνώμη. Βλέπουμε ότι από τα κράτη-μέλη, 20 από αυτά γνωρίζουν το σύστημα αυτό σε διάφορες ε, υπό διάφορε μορφές ε, και υπάρχουν τρόποι να το εισάγουμε αυτό στο ΔΕΚ. Ε, ο λιγότερο επαναστατικό τρόπος ε, θα ήταν απλά να υπάρχει το δικαίωμα να σημειωθεί ότι ένας από τους δικαστές διαφώνησε με την πλειοψηφία χωρίς να αναφέρεται το όνομά του. Αυτό θα ήταν το πρώτο βήμα. Πιο ριζική λύση θα ήταν το δικαίωμα του δικαστή να αναφέρεται το όνομά του στα πρακτικά και ε, κατόπιν έχουμε την πρακτική της δικής μου χώρα, της Δανίας, να έχουμε ε, την ε, εναλλακτική αιτιολόγηση, κάτι που γνωρίζουμε και από το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών και από πολλά άλλα δικαστήρια, όπου τα προβλήματα που αναφέρονται στην έκθεση δεν υπάρχουν. Και τώρα ε, μπορεί να έχουμε κάποιον ο οποίος παρουσιάζει εναλλακτική θέση και δεν υπάρχουν ε, λοιπόν δεν είναι κρυφό ότι υπάρχουν ε, διάφοροι τρόποι να ερμηνεύσει κανείς τον νόμο. Βρίσκω λοιπόν ότι είναι ταπεινωτικό το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να είναι, ένα, να είναι ακόμα το μόνο διεθνές δικαστήριο το οποίο ζει ακόμα στο παρελθόν, δεν δίνουμε την ευκαιρία στους πολίτες μας ε, και τους δικηγόρους ε, ε, τη δυνατότητα να γνωρίζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδόθηκαν οι αποφάσεις αυτές, αλλά να αγνοούμε και την υποχρέωση αυτή για όλα τα θεσμικά όργανα που απορρέουν από τη συνθήκη της Λισαβόνας από το 2009 και μετά είναι υποχρέωση για όλα τα θεσμικά όργανα να διαμορφώσουν μια πολιτική διαφάνεια και το μόνο ε, θεσμικό όργανο που δεν το έχει κάνει αυτό ακόμα είναι, φαίνεται ότι είναι το ΔΕΚ. Κύριε Σκουρή, έχει έρθει η ώρα για ε, αλλαγή. Ε, δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητώ τα ε, κίνητρά σας ε, και γι' αυτό ε, δεν έχετε κι εσείς λόγο να αρνείστε την γνώση αυτών. Ευχαριστώ κύριε Μάση. Νομίζω ότι εμείς ως νομοθέτες δεν αξίζει να χάσουμε ούτε ένα λεπτό για αυτό το θέμα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν θα πρέπει να συζητηθεί σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Γιατί, Γιατί ε, η γνώμη της ε, μειοψηφίας ε, σε μια διάσκεψη κατόπιν της έκδοσης απόφασης, έτσι, μιλούμε, λέμε ότι η γνώμη ενός, δύο, τριών, μιας μειοψηφίας δικαστών τέλος πάντων, ε, ε, ε μπορεί να επηρεάσει την ε, απόφαση, ωραία. Αυτή όμως λαμβάνεται και κλεισμένο των θυρών χωρίς διερμηνία και τελειώνει το θέμα, αλλά η γνώμη της μειοψηφίας την οποία μιλάμε αυτή τη στιγμή ε, εκφράζεται εκ των υστέρων. Στο Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, στον Άτομο Δικαστήριο των ΗΠΑ, η άποψη της ε, μειοψηφίας επέρχεται αργότερα, μετά την έκδοση της απόφασης. Δεν επηρεάζει την απόφαση. Το ίδιο σημαίνει και στο δικαστήριο της Χάγης και σε άλλα δικαστήρια, ακόμα και στο δικά μας στην Ισπανία. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνεται και οι γνώμες της μειοψηφίας, οι γνώμοι ή οι γνώμες της μειοψηφίας δημοσιεύονται αργότερα. Μπορούμε να συζητήσουμε θεωρητικά αυτά τα θέματα ε, στο πλαίσιο μιας συζήτησης συγκριτικού δικαίου κλπ. Αλλά δεν μας αφορούν, άλλωστε δεν εμπίπτουν και στην αρμοδιότητά μας ως νομοθέτη ούτε και αυτή η συζήτηση θα βοηθήσει να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του δικαστηρίου κλπ. Ε, για νομικά θέματα, ακόμα και για το ε, ε φύλλο των αγγέλων, να συζητήσουμε, αλλά όχι στο πλαίσιο της νομοθετικής μας δραστηριότητας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Τάιν. Ναι, ε, πάντα επηρεαζόμαστε πολύ από τις ε, συνθήκες ε, στο δικό μας κράτος μέλος. Εγώ προέρχομαι από κράτος μέλος όπου επιτρέπονται οι διάφανες γνώμες στο συνταγματικό δικαστήριο. Και γι' αυτό προβλέπουμε προβλέψαμε τον κύριο Μέτριο Σμιτ ακριβώς να συζητήσουμε το θέμα των, ε, ε, της πρακτικής αυτής. Καταλαβαίνω όμως ότι δεν συμφωνούν όλοι. Ε, όλοι οι δικαστές με τους οποίους έχω συνομιλήσει και μάλιστα έχω, είχα προσωπικές συναντήσεις με τους δικαστές του δικαστηρίου Ρώτησα ε, δικαστές από την πατρίδα μου και όλοι, όλοι ήταν κατά. Αυτό βέβαια δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Είμαι και εγώ της άποψης ότι Δεν ε, πρέπει να επιβάλλουμε κάτι τέτοιο σε ένα δικαστήριο. Το ίδιο το δικαστήριο γνωρίζει πώς ε, είναι καλύτερο να οργανωθεί και πώς να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και ποια είναι τα προβλήματα. Όσον αφορά το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ε, έχω ασχοληθεί και με αυτό και υπήρξαν περιπτώσεις όπου έχει ασκηθεί πίεση από τα κράτη-μέλη ε, στους δικαστές τους, ιδιαίτερα ε, όταν ε, πρόκειτο για καταδίκη του κράτους μέλους αυτού, πίεση να εκφράσουν οι δικαστές αυτή η διάφωνη γνώμη και μέχρι στιγμής δεν ήξερα ότι σε 7 κράτη-μέλη απαγορεύεται η πρακτική αυτή, αυτό δεν το γνώριζα και ότι στην ε, και μάλιστα στα συνταγματικά δικαστήρια, εκεί που μιλάμε για τα σημαντικά θέματα και όχι για καθημερινά θέματα ερμηνείας περί ανταγωνισμού και τέτοια, ε, Συμφωνώ με τον συνάδελφο Μασίπ ότι είναι προφανώς λάθος στιγμή, δεν έχει ε, νόημα να συνεχίσουμε τις προσπάθειες στο θέμα αυτό. Δεν θα ήθελα να το αποκλείσω τελείως για το μέλλον, αλλά αυτή τη στιγμή μάλλον είναι πολύ νωρίς για κάτι τέτοιο. Μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ πρόημο κάτι τέτοιο. να καταβάλουμε προσπάθειες να εισάγουμε την πρακτική αυτή στο ΔΕΚ. Τα τελευταία δύο χρόνια ε, είχαμε την διαδικασία αυτή, ε, αλλά τελικά καταλήγω σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ, κύριο Σφιέφκα Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που το συζητάμε. Ανεξαρτήτως ε, του αν θεωρούμε πως είναι θεμητό να εκφέρουμε άποψη για το θέμα της με ή όχι. Η κυρία Ραφαέλη μας ε, παρουσίασε μια σύνοψη της κατάστασης στα κράτη-μέλη. Και την ευχαριστώ γιατί έτσι αποκτήσαμε καλύτερη εικόνα της κατάστασης. Απευθυνόμουν στον κύριο Μέσερ Σμιτ, θα ήθελα να πω ότι ε, μερικές φορές ξεχνάμε ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε ένα εθνικό και σε ένα υπερεθνικό δικαστήριο. Σε αυτά τα τελευταία εκδικάζονται υποθέσεις που άπτονται πολλών κρατών. Συνεπώς είναι κάποια διαφορετικά δικαστήρια με ε, διαφορετική σύνθεση. Οπότε δεν θα πρέπει να κρίνουμε το θέμα της δημοσίευσης των, της νόμισης μειοψηφίας με βάση ε, τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε για τα εθνικά δικαστήρια. Το σημαντικό είναι να εξασφαλίσουμε μια ομοιογένεια των αποφάσεων του δικαστηρίου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην συγκεκριμένη περίπτωση και αν δημοσιευόντουσαν οι γνώμες ημιοψηφίας, ίσω κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε εμπόδια στην δημιουργία μια ε, ενιαία νομολογίας. Και θα δίχαζε και τα κράτη-μέλη. Αυτό δεν θα έπρεπε να επηρεάσει το, θέμα, το πώς βλέπουμε το θέμα, αλλά Ε, μην ξεχνάμε και την οικονομική διάσταση. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει προβλήματα καθυστερήσεων εξαιτία του ανεπαρκούς αριθμού δικαστών και αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι η ε, χρηματοδότησή του δεν είναι επαρκής για να προσλάβουν και άλλους δικαστές. Συνεπώς, αν αυξήσουμε το κόστος της μετάφρασης ή της διαρμονίας μπορεί να επηρεάσουμε ακόμα περισσότερο τη λειτουργία του Δικαστήριου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύνεπως, θα πρέπει να τα συζητάμε όλα αυτά βέβαια. Να ξακούσουμε τη γνώμη των δικαστών, των επαγγελματικών, των ακαδημαϊκών και των πολιτικών. Αλλά ας είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τη γνώμη μας. Απευθύνθηκα σε εσά ε, επανειλημμένα και είσαστε ένα ε, από αυτού που γνωρίζουν ε, καλύτερα την κατάσταση. Μπορείτε να μα παρουσιάσετε τη θέση σα. Μια και συζητούμε το θέμα της διαφάνειας, θα ήθελα και εγώ να είμαι όσο πιο ανοιχτός και διαφανής γίνεται, όσο πιο ειλικρινής γίνεται. Γι' αυτό το λόγο ε, να σας πω ότι ε, δεν είμαι υπέρ ούτε και φίλος το, της νόμης της μειοψηφίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να το συζητήσουμε. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το συζητάμε οποτεδήποτε παρουσιαστεί. Όμως, θα ήθελα να περιοριστώ σε ε, ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα. Αν θέλετε να συζητούμε, συζητήσουμε το θέμα της νόμιμης μειοψηφίας, πιστεύω ότι κάτι τέτοιο δεν θα ήταν χρήσιμο για, τις, για τα ολιγομελή τμήματα. Τριμελή, ίσως ούτε και πενταμελή. Ίσως θα μπορούσαμε να, να συζητήσουμε για τις νόμιμες μειοψηφίας στην μείζωνα σύνθεση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι του Γενικού Δικαστηρίου. Α δούμε όμω, και πάλι αν κάτι τέτοιο είναι δυνατό. Όλα βέβαια είναι δυνατά. Αλλά να σας υπενθυμίσω ότι οι κύριες διαδικασίες που έχουμε είναι τα προδικαστικά ερωτήματα, οι προδικαστικές προσφυγές. Ε, οι αποφάσεις που λαμβάνονται εκεί σχετίζονται με την ερμηνεία που δίδει το δικαστήριο απαντώντας σε συγκεκριμένα ερωτήματα που έρχονται από εθνικά δικαστήρια. Δηλαδή τι κάνει το δικαστήριο. Το δικαστήριο ενοποιεί την ερμηνεία. Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι πάντοτε σαφής, διαφανής και ξεκάθαρη. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε ζητείται από το δικαστήριο να ερμηνεύσει σωστά την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Φανταστείτε λοιπόν μια απόφαση του δικαστηρίου με μια απόφαση πλειοψηφία, μια, απόφαση, μια γνώμη πλειοψηφία, μια ε, ε, γνώμη μειοψηφία. Και τι θα κάνει έναντι αυτόν ο Εθνικός Δικαστής, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει την απόφαση του δικαστηρίου. του ζητείτε να ερμηνεύσει το ε, ευρωπαϊκό δίκαιο όπως το ερμήνευσε το δικαστήριο. Οπότε θα αναρωτηθεί τι, πώς ακριβώς το ερμήνευσε το δικαστήριο. Πιστεύω ότι για τέτοιου είδου διαδικασίες το όλο θέμα της ε, γνώμης μειοψηφίας ε, δεν είναι σημαντικό. Ασφαλώς και μπορούμε να το συζητήσουμε. Τώρα, σύγκριση με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εδώ έχουμε κάποια απλά ερωτήματα να απαντήσουμε. Ε, συζητούμε το κατά πόσον αρχές ενός ε, μέλους ε, έχει ή όχι παραβεί ένα από τα 13 άρθρα της Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Της Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και εκεί πράγματι υπάρχουν ε, νόμες και μπορώ να φανταστώ ότι ακόμα και στο δικαστήριό μας, στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις ευθείες προσφυγές ε, έναντι κάποιου κράτους μέλους για παράδειγμα, ε, αν υπάρχει ε, μια ε, ισχυρή γνώμη μειοψηφία, ενδεχομένως θα μπορούσε να δημοσιευθεί γιατί ε, εκεί δεν έχω σημαντικές διαφωνίες ε, αλλά για τα προδικαστικά ερωτήματα που τίθεται θέμα ερμηνείας του νόμου, πιστεύω ότι η δημοσίευση γνώμης μειοψηφία μπορεί να οδηγήσει σε ε, προβλήματα αποδοχής των αποφάσεων του δικαστηρίου και με εξέπληξε που άκουσα ότι ε, η αν μια απόφαση είναι απόφαση πλειοψηφίας δεν έχει ε, πλήρη εφαρμογή ε, και κύρος. Δεν είναι δημοκρατικό αυτό. Στη δημοκρατία η πλειοψηφία είναι πλειοψηφία. Και αν η πλειοψηφία εκφραστεί έχει το ίδιο κύρος ε, με την ομοφωνία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Δεν νομίζω ότι χωρά Χωρεί αμφιβολία. Δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι μια απόφαση δικαστηρίου είναι, έχει λιγότερο κύρος επειδή δεν συμφώνησαν όλοι οι δικαστές. Αυτό πρώτη φορά το ακούω ως επιχείρημα. Αν αυτό είναι το σκεπτικό για την δημοσίευση της συγγνώμης μειοψηφία, εγώ θα έλεγα το ακριβώς αντίθετο. σα ευχαριστώ. Ο κύριος Μέσερσμιτ θέλει να μιλήσει. Πρέπει να διευκρινίσουμε ένα στοιχείο δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο ο οποίος θα επιβάλλει σε οποιονδήποτε δικαστή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να εκδώσει μία μειοψηφούσα ή διαφωνούσα γνώμη. Αυτό που θέλουμε να δώσουμε είναι τη δυνατότητα, την εναλλακτική λύση να δώσει μία μειοψηφούσα άποψη. Εάν όλοι οι δικαστές συμφωνούν, τότε δεν θα υπάρχει μια ψηφούσα γνώμη. Αυτό όμω που συζητούμε εμείς μπορεί να είναι υποθετική κατάσταση, δεν είναι υποθετική, αλλά μια πραγματική κατάσταση ένας δικαστής διαφωνεί με την πλειοψηφία. Και αυτός ο δικαστής του διαφωνών θα έχει το δικαίωμα να εκφράσει την διαφωνούσα γνώμη. Ε, στη μειοψηφία που βρίσκεται, νομίζω ότι οποιοδήποτε ευρωπαϊκό ίδρυμα ή φορέας ή θεσμικό όργανο θα ήταν ανάστατο και αγανακτισμένο αν δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Σκεφτείτε, εάν ε, η Κομισιόν έλεγε ή το Κοινοβούλιο έλεγε ότι εμείς δεν θέλουμε διαφάνεια διότι δεν μας αρέσει, δεν θέλουμε να ξέρει κανείς ποιος ήταν ο διαφωνών ή ο μειοψηφών, αλλά στο σύγχρονο κόσμο έχουμε την ε, υποχρέωση και οι συνθήκες ε, και εσείς κύριε Σκουρή επιβάλλουν να ακολουθήσουμε τη συνθήκη και αν δεν δίνεται αυτή η πιθανότητα, ε, τότε νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν είναι ε, ικανό να επιτελέσει το καθήκον του. Έχω διαβάσει εκατοντάδες αποφάσεις ε, στο Ευρωπαϊκό του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και δεν διαβλέπω ότι αποκλίνουν ή διαφέρουν από τις αποφάσεις τις εθνικές στη Δανία. Τώρα, θα πρέπει να δώσουμε, πιστεύω, τη δυνατότητα στη σε μία μειοψηφία να εκφραστεί. Σκεφτείτε την ηρωνική κατάσταση όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, ε, ε, ε, το, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, άρθρο 6, υπάρχει διαφωνία. Υπάρχει διαφωνία σε μία δίκη. Και από το Στρασβούργο έρχεται μία διαφωνούσα γνώμη και μια άλλη άποψη από το Λουξεμβούργο, ε, μια άλλη απόφαση επί του άρθρου 6 χωρίς διαφωνούσα γνώμη. Λοιπόν, μια απόφαση από το Στρασβούργο έχει διαφωνούσα, μια άλλη από το Λουξεμβούργο δεν έχει. Πώς θα μπορέσετε εσείς σε μια τέτοια δικογραφία, ας πούμε, ε, όπου υπάρχουν διαφορετικές απόψεις να αρνηθείτε την υποθετική περίπτωση όπου ένας μειοψηφών συνάδελφος ε, δεν έχει το δικαίωμα να εκφράσει την μειοψηφούσα γνώμη του. Εντάξει, δέχομαι το επιχείρημα ότι αυτό δεν είναι δυνατόν σε μία ε, μικρή δικαστική ομάδα, τριών δικαστών ας πούμε, αλλά αν πούμε στην ολομέλεια του δικαστηρίου, γιατί δεν είναι δυνατόν, γιατί δεν... Ε, ε, γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Επειδή δεν λειτουργεί στις προδικαστικές αποφάσεις, επειδή δεν λειτουργεί σε ένα μικρό δικαστικό σώμα περιορισμένο, αυτό είναι το βασικό επιχείρημα που θα μας απαγορεύσει σε άλλων μειοψηφών ε, δικαστή να εκφράσει την άποψή του παντού και πάντοτε. Δεν το πιστεύω αυτό, δεν συμφωνώ. Η Πρόεδρος, κοιτάξτε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν είναι το δικαστήριο του κυρίου Σκουρί, είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όλων μας. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον πρόεδρό του να απαντήσει. Ο κύριος Σκουρής, είπα τι ήθελα να πω. Μερικές φορές πρέπει να διαφωνούμε. Η διαφωνία είναι και αυτή ε, με στη ζωή. Είναι φυσιολογικό. Όσον αφορά εμένα, εγώ είμαι σταθερός στις απόψεις. Εμένα στην άποψή μου που εξέφρασα όσον αφορά την αναγκαιότητα, μη αναγκαιότητα των separate opinions. Ίσως κύριε Μέσσεσμιτ, εμένα μου αρέσει να ζω περισσότερο στο παρελθόν. Ευχαριστώ πολύ λέει η Πρόεδρος. Το τρίτο μέρος της ακρόασής μας και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Βέσνα Νάγκλιτς από το τμήμα γάμα το τρίτο τμήμα της ε, πολιτικών υποθέσεων να μας παρουσιάσει την άποψή της για τις εθνικές πρακτικές όσον αφορά την προσβασιμότητα ε, των, σε δικογραφίες, στα έγγραφα των δικαστηρίων. Σε δικόγραφα. Και ε, θα ήθελα ε, να παρακαλέσω τους επόμενους ομιλητές που δεν φταίνε βέβαια σε τίποτα να είναι σύντομοι, να είναι σύντομοι. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε τη δυνατότητα να παρουσιάσω τη μελέτη αυτή. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη αλλά και ε, να γίνω κατανοητή. Τι, ποιο είναι λοιπόν το θέμα της ε, ε, μελέτης αυτής. Ε, μιλάμε για την πρόσβαση τρίτων σε έγγραφα του δικαστηρίου. Μπορεί λοιπόν κάποιος τρίτος να έχει πρόσβαση ε, σε έγγραφα του δικαστηρίου, είναι δηλαδή εμπιστευτικά τα έγγραφα αυτά ή κάποιες πτυχές του και δεύτερον πώς η προσπάθεια απαιτείται από το, τους τρίτους αυτούς για να έχουν πρόσβαση σε κάποια έγγραφα. Αρκεί να στείλει ένα email στο προσωπικό κάποιου δικαστηρίου και να πει ότι θα ήθελα παρακαλώ πρόσβαση στην ε, υπόθεση Χ. Είναι απαραίτητο να προσέλθει ε, προσωπικά στο δικαστήριο για να λάβει αντίγραφο. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να καταλάβουμε γιατί ανατέθηκε η μελέτη αυτή. Ένας από τους λόγους ήταν ότι η Επιτροπή Τζούρι πέρσι ότι ήρθαν σε επαφή με την Επιτροπή Τζούρι κάποιοι ε, νομικοί οι οποίοι είπαν ότι δεν καταλαβαίνουμε γιατί υπάρχουν ε, δυσκολίες να λάβουμε ένα έγγραφο από ε, ένα δικαστήριο το οποίο είναι διαθέσιμο ε, σε κάποια βάση μητρώου του κράτου μέλους. Εάν όμως προσφύγω στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν, όπου υπάρχει το έγγραφο σε μια γλώσσα που καταλαβαίνω δεν μπορώ να έχω πρόσβαση επειδή θεωρείται εμπιστευτικό οι νομικοί που ήταν παρόντες σε μια κροματική διαδικασία και που έχουν λάβει τα πρακτικά της ε, διαδικασίας αυτής, ε, για παράδειγμα στα Ουγγρικά, ε, γνωρίζοντας ότι υπάρχει το έγγραφο αυτό στα γαλλικά, όταν ζήτησαν από το δικαστήριο το έγγραφο αυτό στα γαλλικά, δεν τους δόθηκε, διότι και πάλι το δικαστήριο απάντησε ότι πρόκειται για έγγραφο εσωτερικής κυκλοφορίας και δεν επιτρέπεται να παραδοθεί στον ενδιαφερόμενο. Όσον αφορά λοιπόν ε, την πρόσβαση, ε, ποια είναι η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον κόσμο γενικά. Γενικά, ε, ο δικαστικός τομέας εξαιρείται από την πρόσβαση αυτή σε δημοσία έγγραφα που ισχύει. Έτσι λοιπόν είναι δυνατόν οι γιατροί τους ε, να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα που έχουν να κάνουν με την ε, διοικητική πλευρά. Ή αν ε, δεν εξαιρείται ο δικαστικός τομέας, σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν εξαιρέσεις που σχετίζονται με τις συζητήσεις του δικαστηρίου, κάποιοι τύποι κάποιους τύπους ε, εγγράφων. Ε, έτσι λοιπόν είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς ότι υπάρχει πρόσβαση τρίτων σε αρχεία του δικαστηρίου. Και εάν δεν ισχύει αυτό και πάλι μιλάμε για κάποιο δικαίωμα πρόσβασης ε, στα δικαστικά έγγραφα, τότε μπορεί Τρίτη, να έχουν πρόσβαση στα αρχεία μόνο εφόσον κλείσουν ε, και όχι όσο εκκρεμεί ακόμα υπόθεση στο δικαστήριο. Πολύ σύντομα λοιπόν να απαντήσω ποια είναι η κατάσταση. Αν δούμε την κατάσταση αυτή τη στιγμή, πρέπει να πούμε ότι ε, δεν υπάρχουν πολλές χώρες στον κόσμο που να παρέχουν ε, ανοιχτή πρόσβαση σε τρίτους ε, στα αρχεία των δικαστηρίων. Εάν όμως δούμε το θέμα αυτό πιο δυναμικά, στο χρόνο δηλαδή, και πάμε πίσω 40-50 χρόνια, θα παρατηρήσουμε το εξής πολλά κράτη αποφάσισαν να υιοθετήσουν νομοθεσία σχετικά με την πρόσβαση ε, σε ε, δημόσιες πληροφορίες και με την έλευση του διαδικτύου. Ε, οι δημόσιες αρχές έχουν αποφασίσει να δώσουν περισσότερη πρόσβαση. Η τάση λοιπόν αυτή που θεωρούμε ότι είναι σημαντική όχι μόνο για το νομοθετική κυβέρνηση, αλλά και για το δικαστικό τομέα, τότε μάλλον υπάρχει μια τάση που να υποχρεώνει το δικαστικό τομέα να είναι όσο γίνεται πιο ανοιχτός. Στην ε, παρουσίασή μου θα ε, επικεντρωθώ στον Καναδά που δεν είναι κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί ε, στον Καναδά, διότι φαίνεται ότι το δικαστικό του σύστημα μπόρεσε να αντιμετωπίσει κάποια πολύ προβληματικά σημεία. ο Καναδάς έχει την προσέγγιση της ανοιχτής πρόσβασης. Υπάρχει συνταγματική αρχή ότι πρώτον ε, ο καθένας μπορεί να πάει σε ένα δικαστήριο και να είναι παρόν κατά την ακροματική διαδικασία και δεύτερον οποιοδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση στα έγγραφα υπό τους όρους που ισχύουν για το δικαστήριο αυτό. μάλλον συγγνώμη, επιτόπου στο δικαστήριο. Βέβαια, ο κανόνα αυτό είναι ξεπερασμένο στη στιγμή που όλοι έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και έτσι εξέτασαν πώ μπορούν να ε, υιοθετήσουν τι ε, νέε τεχνολογίε και να δώσουν πρόσβαση στα δικαστικά έγγραφα σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο. Ένα από τα πιο προβληματικά θέματα είναι η πρόσβαση από τρίτους εξ αποστάσεως, ε, διότι τίθεται θέμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων και ο Καναδάς είπε ότι αυτό μπορούμε να το λύσουμε ε, υποχρεώνοντας ε, τους ε, αντιδίκους ε, και τους δικηγόρους τους να γνωρίζουν ότι οποιοδήποτε έγγραφο μπορεί να το δει κάποιος τρίτος. Έτσι λοιπόν είναι δική τους ευθύνη αν συμπεριλάβουν υπερβολικές πληροφορίες, κάτι που να είναι άσχετο με την δικαστική εξέταση. Το καναδικό σύστημα είναι επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον διότι η πρόσβαση εξ αποστάσεως είναι υποχρεωτική. Δηλαδή δεν είναι... Δεν αρκεί το δικαστήριο να πει ότι, ότι ναι μπορείτε να έχετε πρόσβαση αλλά θα πρέπει να ε, ε, έρθετε προσωπικά. Ε, είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πρόσβαση εξ Ο τρίτος επίσης πρέπει να γνωρίζει ποια είναι τα δικαιώματά του και ε, ποιες είναι οι υποχρεώσεις του. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιος μηχανισμός ελέγχου ώστε να μην δίδεται πρόσβαση σε πρόσωπα που μπορεί να καταχραστούν του δικαιώματος ε, της πρόσβασης ε, σε διαφόρων τύπων πληροφορίες. Δυστυχώς δεν μπορώ να πω σε λεπτομέρειες λόγω της πίεσης του χρόνου. Επίσης, ε, ο καναδικός ε, δικαστικός ε, τομέας γνωρίζει ότι δεν αρκεί απλά το να δίνει ακατέργαστα δεδομένα. Κάθε δικαστήριο, λοιπόν, έχει παρέχει τις λειτουργίες αναζήτησης διότι τα κατάρτιστα δεδομένα μπορεί να μην έχουν πολύ νόημα, θα πρέπει να μπορεί κανείς ε, να κατηγοριοποιήσει τα δεδομένα, ώστε να μπορέσει να εξάγει τις πληροφορίες που αναζητά. Ε, όσον αφορά το δικαστήριο, λοιπόν, ε, είναι προσβάσιμες ε, οι ε, αποφάσεις του δικαστηρίου, όχι όμως ε, τα εσωτερικά έγγραφα. Και όσον αφορά την πρόσβαση σε συγκεκριμένα αρχεία, οποιοδήποτε τρίτος θέλει να λάβει ένα έγγραφο θα πρέπει καταρχήν να απευθυνθεί στην γραμματεία του δικαστηρίου που κατόπιν ε, θα ζητήσει την άδεια από το αρμόδιο τμήμα και αν δεν δοθεί η άδεια τότε ο τρίτος δεν έχει δικαίωμα πρόσβαση στο συγκεκριμένο έγγραφο. Η διαδικασία αυτή είναι πολύ χρονοβόρα και επαχθής και ε, εξετάζοντάς το υπό ε, το φως της ε, καναδικής διαδικασίας μπορούμε να αμφισβητήσουμε αν είναι λογικό να συνεχίσουμε με την πρακτική αυτή. Θα κλείσω την παρουσίασή μου τώρα διότι ο κύριος Πάτσερ Τζόις θα μας παρουσιάσει τις δικές του προσωπικές εμπειρίες όσον αφορά την πρόσβαση σε έγγραφα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Πάτσερ Τζόις, να ευχαριστήσω και να αποχαιρετήσω τον κύριο Σκουρί. Πιστεύω ότι αυτός ο διάλογος και η ανταλλαγή απόψεων με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την νομοθετική μας εργασία. Και θα έλεγα ότι ευχόμαστε όλοι να συνεχιστεί αυτή η στενή συνεργασία. Και τώρα δίνω στον κύριο Πράτσετ Τζόις, ο οποίος είναι μπάριστερ και μιλάει εκτός μικροφώνου δυστυχώς. Εκτός μικροφώνου ο μιλητής. Sorry. Αγαπητά μέλη, κυρία Πρόεδρε, θα ήμουν πολύ σύντομο. Έχω ε, ορισμένε σημειώσει που θα δημοσιευθούν αργότερα. Η πρώτη παράγραφος των σημειώσεων μου εκφράζει τις ευχαριστίες μου για την πρόσκληση. Η δεύτερη αναγνωρίζει την πολύτιμη εργασία την οποία έχει κάνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τα τελευταία 60 χρόνια. Και αυτές οι δύο παράγραφοι πιστεύω ότι μπορούν να μπουν στα πρακτικά. Το θέμα είναι ευρύο, ευρύτατο, αλλά η δική μου πρόσκληση είναι συγκεκριμένη όσον αφορά την ουσία του θέματος που είναι πρόσβαση σε, στις δικογραφίες αλλά και ως επαγγελματίας του κλάδου ε, ως επαγγελματίας, ως μπάριστερ λοιπόν, είμαι υποχρεωμένος και έχω καθήκοντα έναντι και των δικαστηρίων, των δικαστών και των πελατών μου. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαι σε θέση να ερευνήσω την υπάρχουσα νομολογία ε, ε, ε, εμπεριστατωμένα, να την εφαρμόσω και να την παρουσιάσω. Υπάρχουν λοιπόν πέντε στάδια στην εργασία μου. Κατά πρώτον να κατανοήσω τον νόμο, την νομοθεσία. Δεύτερον, να παράσχω τις σωστές νομικές συμβουλές στους πελάτες μου. Τρίτον, να είμαι σε θέση να επιχειρηματολογήσω την υπόθεση αυτή ενώπιον του δικαστηρίου. Να είμαι σε εσύ να παρουσιάσω με σαφήνεια την υπόθεση και πέμπτον να ε, φροντίσω να παρασχεθεί όλη η αναγκαία υποστήριξη στο δικαστήριο. Είχα το πλεονέκτημα και την τιμή να διαβάσω την ε, μελέτη της κυρίας Ναγκλίτς και τη διάβασα με μεγάλο ενδιαφέρον. Εάν μου επιτρέπετε να πω, η μελέτη αυτή προσφέρει μία λεπτομερή, ουσιαστική και ολοκληρωμένη ανάλυση των προβλημάτων των σημαντικών προβλημάτων που ε, αφορούν στην ε, πρόσβαση ε, στις δικογραφίες. Για να σας πω λοιπόν τώρα πώς και βρέθηκα εδώ. Όταν πήγα στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου πέρσι το Μάρτιο, όχι για να εξασκήσω το επάγγελμά μου, αλλά ως παρατηρητής. Δηλαδή ουσιαστικά ήμουν ένα τρίτο μέρος στη διαδικασία αυτή, κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων της υπόθεσης από τους ε, συναδέλφους αναφέρθηκαν, πήρα διάφορες ε, σημειώσεις και παρέπεμπαν, παρέπεμπαν οι συνάδελφοί μου σε συγκεκριμένα άρθρα και παραγράφους ε, που τις ε, γνώριζαν σαφέστατα και οι συνάδελφοί μου δικηγόροι και οι δικαστές. Αλλά για κάποιον, σαν και εμένα, που ήμουνα τρίτο μέρος, εκτός δηλαδή των, εσωτερικών διαδικασιών του δικαστηρίου, οι παρουσιάσεις αυτές και οι εισηγήσει ήταν άνευ νοήματος. Θα μπορούσε να ήταν και στα κινέζικα δηλαδή. Δεν μπορούσα να τις κατανοήσω. Μου φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει ένα έλλειμμα ενημέρωση, ένα έλλειμμα, έλλειμμα πληροφόρησης, τουλάχιστον όσον αφορά τους επαγγελματίες παρατηρητές των διαδικασιών. Όταν ζήτησα τα έγγραφα, τις δικογραφίες μου είπαν ότι δεν μπορούν να μου τα δώσουν διότι δεν έχω πρόσβαση, αποκλείομαι από την πρόσβαση στη δικογραφία για να διατηρηθεί το κύρος του δικαστηρίου παρόλο που το περιεχόμενο της δικογραφίας ε, συνά, τότε ήταν σύμφωνα με τις υποθέσεις που χειριζόμουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και εφόσον λοιπόν δεν μπόρεσα να λάβω τα έγγραφα της δικογραφίας, δεν μπόρεσα και ενημερώσω, να ενημερώσω τις δικές μου εθνικές αρχές για την, τις υποθέσεις αυτές. Ε, ενώ ήμουν επίσημος παρατηρητής. Έτσι λοιπόν ε, μου δημιουργήθηκαν διάφορες επιφυλάξεις. Πρώτον, όσον αφορά την απονομή δικαιοσύνης, αλλά δεύτερον και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα, η οποία για μένα είναι απαραίτητα ως επαγγελματίες. Μου φαίνεται ότι όλη αυτή η ιστορία της πρόσβασης στα δικόγραφα είναι φορτωμένη, υπερβολικά φορτισμένη με υπέρ και κατά απόψεις. Αυτό που θέλω να πω ουσιαστικά είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα μπορούσε να είναι πιο ανοιχτό, πιο διαφανές και να προωθήσει καλύτερα την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Εάν το έπρατε αυτό το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν θα υπονόμευε ούτε θα διακύβευε την ακαιρεότητα και το κύρος του αλλά θα βελτίωνε την προσβασιμότητα και την κατανόηση. Και αυτό θα επέφερε και μια καλύτερη θετική γνώμη των πολιτών. Προσπάθησα λοιπόν να εξετάσω και τις, να, να καταγράψω και τις απόψεις άλλων που συμμετείχαν στη διαδικασία και ήταν στην ακρόαση. Όπως Λοιπόν, ήδη ελέγχθη, έχοντας υπόψη τους νέους διαδικαστικούς κανονισμούς, η έκθεση για την ακρόαση στην οποία πήγα εγώ και στις άλλες ακρεώσεις δεν θα δημοσιευθεί καθόλου. Τα πρακτικά, τα πρακτικά δεν θα δημοσιεύονται καθόλου πουθενά. Πιστεύω ότι αυτό είναι μια μεγάλη επιστοδρόμηση. Και αυτό στο, στην παράγραφο 6.3 τελεία 2 αναφέρεται στην, ε, ναι, στην μελέτη της κυρίας Νάγκλιτς. Πράγματι είναι μια μεγάλη επιστοδρόμηση αυτή η απαγόρευση. Και τέλος, ε, στη συνέχεια αυτών που είπε η κυρία Μαγκάουεν, θα πρέπει να υπάρχει μία επιτροπή πλήρως ενημερωμένη και αξιο, αξιόπιστη, ε, η οποία θα είναι αρμόδια για τις διαδικασίες, ενημέρωση διαδικασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή στην οποία να μπορούμε εμείς να προσφεύγουμε για ενημέρωση και πληροφόρηση. Αυτά είχα να πω, κύριε Πρόεδρε. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κέλλερτ. Ο κύριος Κέλλερτ από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θέλει να παρέμβει. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα σας δώσω πολλές πληροφορίες. Θέλω απλώς να σας πω ότι είναι ένα σημαντικό θέμα για το δικαστήριο η έκθεση της κυρίας Νάγκλητς. αποδεικνύει ότι η κατάσταση στα διαφορετικά κράτη-μέλη η κατάσταση στα κρατη διαφέρει. Είναι ένα θέμα που εξελίσσεται. Εμείς το συζητάμε εσωτερικά. Θα ήθελα απλώς να σας ενημερώσω για το ε, report for the hearing. Ε, ε, η έκθεση αυτή δεν υπάρχει πια, όχι ότι δεν θα δημοσιεύεται. Δεν υπάρχει για ένα πολύ απλό λόγο. και το δικαστήριο πρέπει να κάνει περικοπές. Οπότε θα πρέπει να περιοριστούμε σε αυτά που είναι απολύτως απαραίτητα για την σωστή απονομή της δικαιοσύνης. Είναι χρήσιμη η έκθεση ε, της ε, κροματικής διαδικασίας, αλλά απαιτεί χρόνο ε, από τους δικαστές, απαιτεί χρήματα για τη μετάφραση, ε, πέραν του γεγονότος ότι αυτή η έκθεση ε, δεν υπάρχει σε άλλες σε νομικές τάξεις. Οπότε χρειάστηκε να κάνουν περικοπές και επιλέξαμε αυτό, μεταξύ άλλων. Μην ξεχνάτε ότι ε, έχουμε περιορισμένους πόρους. Τα μέτρα λιτότητας μας επηρεάζουν και εμάς. Δεν είναι θέμα έλλειψης επιθυμίας να δημοσιεύσουμε ένα έγγραφο. Δεν υπάρχει πλέον αυτό το έγγραφο. Ευχαριστώ. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνουμε την ε, ακρόαση αυτή και ευχαριστώ όλους όσους ε, συμμετείχαν στην ακρόαση και έξω ε, έχετε όλα τα έγγραφα των ε, ομιλιών όσα υπάρχουν, όσα διατίθενται και ευχαριστώ ιδιαίτερα το Policy Department, ε, το αρμόδιο τμήμα, το οποίο βοήθησε στη διοργάνωση της ακρόσης αυτής και πιστεύω ότι όλοι εμπλουτιστήκαμε με πολλές γνώσεις και ευχόμαστε, κάθε επιτυχία στην ολοκλήρωση της έκθεσης ε, στην κυρία Τάιν. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους συμμετάσχοντες και όσους έρχονται από τους επαγγελματικούς κλάδους και μας έδωσαν μια πολύ ζωντανή εικόνα της, ε, του θέματος. Δεν θα προχωρήσουμε τώρα στο επόμενο θέμα, όπως σας είπα. αλλά όπως σας είπα στην αρχή θα συζητήσουμε τα αποτελέσματα της συνάντησης των συντονιστών που έγινε στο Στρασβούργο και η οποία ήταν πολύ ε, πλούσια σε θέματα. Καταρχάς, λοιπόν, ο ορισμός των εισηγητών ή αυτών που θα συντάξουν τις γνωμοδοτήσεις. Η κυρία Λίχτεμπεργκερ για την ε, ασυλία του κυρίου Αλεξάνδρου Αλβάρο. Δε, δεύτερος εισηγητής ο κύριος Καρίμ για την 19η έκθεση του Better Lawmaking 2011. Τρίτον, ο κύριος Μπόρες εισηγητής για την WIPO, η κυρία Γκέριγκερ για, την, για το cloud computing ε, στην Ευρώπη, ο κύριος Λόπεζ εισηγητής και τα λέω στα γαλλικά. Sur l'appartenance à l'Union européenne de la sécession d'un territoire d'un État membre. c'est un Also, der Sezession ε, απόσχεση όσον αφορά τις επιπτώσεις για την απόσχεση της, ε, ε, του εδάφους ενός της κάποιου τμήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν συνεχεία, εισήγηση για ε, την είσοδο τρίτων υπηκών, υπηκών τρίτων χωρών για σκοπούς έρευνας, ε, θελοντική υπηρεσία κλπ. Ο κύριος Στογιάνοφ θα είναι αρμόδιος, θα είναι ο συγητής και τέλος η, α, ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και μελέτη των τροπολογιών. Εδώ δεν πρόκειται για ε, τυπική επίσημη ε, γνωμοδότηση, αλλά λόγω χρονικής πίεσης θα παρουσιαστούν οι τροπολογίες εξονόματος του κυρίου Λένα και μου και θα ψηφιστούν άμεσα και θα παραπενθούν στην ε, ε, αρμόδια επιτροπή και το επόμενο θέμα είναι η προφορική ερώτηση για την του, πρόοδο του προγράμματος Στοκχόλμης μαζί με την Επιτροπή Λίμπε και ΑΦΚΟ. Ε, κοινή ε, προφορική ερώτηση το Μάιο στο Στρασβούργο. Κοινή προφορική ερώτηση Μάιο Στρασβούργο. Επόμενο θέμα, η Επιτροπή μας ε, θα ζητήσει εντολή για μία έκθεση του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαιοσύνης Scoreboard. Εν συνεχεία, η επόμενη Προεδρία της Λιθουανίας στη συνεδρίαση της ομάδας της 9 Ιουλίου θα παρουσιάσει τις προτεραιότητές της και ε, αυτό θα γίνει από τον Υπουργό κ. Μπερνατώνης και τον Υπουργό Πολιτισμού κ. Μπυρώτης στις 8 Ιουλίου θα υπάρχει μια έκτακτη ε, συνάντηση μισής ημέρας της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων, εξαιρετική συνεδρία, στις 8 Ιουλίου, το απόγευμα, το απόγευμα. Μισή μέρα μόνο έκτακτη συνεδρίαση για να μπορέσουμε να διευθετήσουμε το πρόγραμμά μας. Και τέλος, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Επίτροπος κ. Σεφτκοβιτς, στις 19 Ιουνίου θα έρθει σε εμά να μιλήσει για την πρόοδο του διοικητικού δικαίου. Α, της διοικητικής διαδικασίας. Τέλος, ε, την, στην επόμενη Ολομέλεια στο Στρασβούργο θα υπάρχει η δυνατότητα να επισκεφθούμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όσα μέλη της Επιτροπής μας ενδιαφέροντες να συμμετάσχουν σε αυτό, παρακαλώ να ανακοινώσουν την πρόθεση, την επιθυμία τους στη γραμματεία. Και Έχουμε και μια διακοινοβουλευτική συνάντηση για το πρόγραμμα στο Χόλμης μαζί με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ στις 20 Ιουνίου. Για το θέμα δια... στο copyright, για αυτούς που έχουν προβλήματα όρασης, θα υπάρξει προφορική ερώτηση στην Ολομέλεια του Μαΐου, Στρασβούργο. Και τι άλλο έχουμε. Οι συντονιστές αποφάσισαν όσον αφορά τον προϋπολογισμό του 2013 να υπάρχει μία γνωμοδότηση, δηλαδή να δοθεί εντολή για σχέδιο έκθεσης Α, για εισηγητή επί του σχεδίου προπολογισμού της Κομισιόν συγκεκριμένα στα θέματα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Να υπάρξει εισήγηση δηλαδή επ' αυτού. Επίσης, η, ε, η Επιτροπή μας ε, όσον αφορά τη νομική βάση και στο θέμα της διάκρισης του φύλου και της ίσης κατανομής των φύλων στη νομική βάση αυτού του θέματος θα συντάξει μία γνωμοδότηση. Η ψηφοφορία δεν θα γίνει σε αυτή τη συνεδρία, αλλά στην επόμενη. Τέλος, υπάρχει ακόμα το θέμα της επίσημης αντιπροσωπείας Επιτροπής μας στις 17 και 18 Ιουλίου, που θα πάμε στη Λιθουανία για να συναντήσουμε τους επίσημους εκπροσώπους στο Βίλνιους και να συζητήσουμε την προτεραιότητα της Προεδρίας. Και τέλος, και εδώ φτάνω στο τέλος, όσον αφορά τους συντονιστές στο Στρασβούργο, η Επιτροπή μας, η Γιούρη, μαζί με την Επιτροπή Αναφορών, μας ζητήθηκε να οργανώσουμε ένα hearing, μία ακρόαση με θέμα των Ευρωπαίο, τον ε, ε, ε, το διαμεσολαβητή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έτσι μπορούμε και προχωρούμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης που είναι η ηλεκτρονική ταυτοποίηση. Ηλεκτρονική και υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην ιστορική αγορά. Ο κύριος Μεζαρός έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν την παρουσίαση του σχεδίου γνωμοδότησης θα παρακαλούσα να μου επιτρέψετε να εκφράσω τους αρμόδιους ε, της Επιτροπής Γιούρη και τη ε, Γραμματεία για την εξαιρετική του συνεργασία κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες. Επιτρέψτε μου τώρα να αναπτυχθώ πάνω στις, ε, να, να αναπτύξω τις βασικές αρχές της νομοδότησης ε, Γιούρη σχετικά με κανονισμό του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνη για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Ε, τα θέματα αυτά ενδιαφέρουν και ε, επιχειρήσεις και ε, ιδιώτες και γι' αυτό επικροτώ την πρόταση της Κομισιόν για, σχετική, για τα θέματα αυτά είναι η τελευταία από τις 12 δράσεις ε, κλειδιά που προτείνονται στην ε, πράξη για την ενιαία αγορά και ανταποκρίνεται στις ανάγκες ε, των των στην ψηφιακή αγορά για να διασφαλίσει ένα συνεχτικό νομικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές σε ευρωπαϊκό, συναλλαγές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, στόχος είναι να, να διασφαλίσουμε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να μπορούν να χρησιμοποιούν τα προγράμματα αυτά για ε, πρόσβαση σε ε, δημόσιες υπηρεσίες σε άλλα κράτη-μέλη όπου ήδη υπάρχουν τέτοια, προγράμματα. Ο κανονισμός απαιτεί αμοιβαία αναγνώριση ανάμεσα σε διάφορα εθνικά συστήματα ευρωπαϊκής, ε, ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Πιστεύω ότι οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι εθνικές αρχές χρειάζονται ε, μια αξιόπιστη ψηφιακή εσωτερική αγορά για την δουλειά τους, για τις σπουδές τους, για τα ταξίδια τους και διάφορες άλλες δραστηριότητες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή με κάποιες εξαιρέσεις οι κυβερνήσεις των κρατών μελών ε, παρέχουν υπηρεσίες επαχθής, ε, δεν τις παρέχουν ηλεκτρονικά ή τις ε, παρέχουν σε περιορισμένο τόπο και χρόνο και μάλιστα ενίοτε με υψηλότερο κόστος. Ποια είναι τα ωφέλη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διασυνοριακές περιπτώσεις. Καταρχήν, οι συναλλαγές αυτές ε, είναι πιο βολικές, ε, εξοικονομούν χρόνο και κόστος από ότι είναι οι προσωπικές ε, συναλλαγές με τις κυβερνήσεις. Ο κανονισμός θα έχει θετικό αντίκτυπο στους εξής τομείς. Τις ηλεκτρονικές συμβάσεις, την εκπαίδευση και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες. Διασφαλίζει νομική ασφάλεια στην περίπτωση της ε, χρήσης ηλεκτρονικής ε, ταυτοποίησης ε, εντός της εσωτερικής αγοράς. Ως εισηγητής τη γνωμοδότηση της Γιούρη θα ήθελα να τονίσω ότι η νομική βεβαιότητα θα πρέπει να διασφαλίζεται με τον νέο κανονισμό ώστε οι επιχειρήσεις και οι πολίτες να μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στις διασυνοριακές ηλεκτρονικές συναλλαγές και γι' αυτό προτείνω κάποιες τροποποιήσεις ε, στην ε, διαδικασία κοινοποίησης ε, και κάποιες διευκρινήσεις όσον αφορά τη ευθύνη και την προστασία των δεδομένων. Ταυτόχρονα, η περιττή γραφειοκρατία και τα περίτα άχθη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να αποφευθούν. Τέλος, προτείνω μια σειρά τροποποιήσεων ε, όσον αφορά την εφαρμογή των ε, πράξεων κατουσιοδότηση όπως προτείνονται από την Επιτροπή, ώστε να αντικατοπτρίζονται καλύτερα οι στόχοι των άρθρων 290 και 291 της ε, Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα, σε μια σειρά θεμάτων, δεν μας φαίνεται ε, ε, ότι αντίθεται η ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις ε, χρειάζεται περισσότερη διευθύνση σχετικά με το περιεχόμενο της ανάθεσης αρμοδιοτήτων. Έχουν υποβληθεί 40 περίπου τροπολογίες. Από ό,τι γνωρίζω, η προθεσμία για περαιτέρω υποβολή τροπολογιών από τους συναδέλφους είναι 15 Μαΐου 2013. Σας ευχαριστώ πολύ. Dankeschön. Äh, möchte sich jemand zu κάποιος άλλος να μιλήσει. Δεν νομίζω, τα είπαμε όλα. 15 Μαΐου προθεσμία τροπολογιών. Α, η κυρία Τέλερ. Sorry, as shadow I forgot. Ε, Ευχαριστώ τον εισηγητή για την έκθεσή του. ορίζω την πρωτοβουλία της Κομισιόν. Είναι ένα σημαντικό τμήμα της ψηφιακής ατζέντα. Η σημερινή νομοθεσία είναι πεπαλαιωμένη. Από την άλλη μεριά το περιβάλλον είναι πολύ ε, ποικίλο. Τα κρατη έχουν διαφορετικά συστήματα. Ε, μια, αυτή η πρωτοβουλία θα βοηθήσει και τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Χρειαζόμαστε εναρμόνιση ε, στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, αλλά αυτό βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Ε, πρέπει να βελτιώσουμε τις, την εμπιστοσύνη με την αποδοχή των νέων προτάσεων αλλά και με τη βελτίωση νομικής ασφάλειας. Ορισμένα σημεία της πρότασης δημιουργούν σύγχυση για το πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη. Για παράδειγμα, όροι για την κοινοποίηση συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Απαιτείται ε, από τα κράτη-μέλη να γίνεται ε, ε, μονοσήμαντη χορήγηση ηλεκτρονικών στοιχείων σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Αυτό όμως είναι ασαφές. Απ' την άλλη μεριά έχουμε τις ε, ε και εκτελεστικές πράξεις προτείνει η Κομισιόν. Ορισμένα από αυτά θα πρέπει να ξεκαθαριστούν ή ορισμένες αυτές τις πράξεις δεν φαίνονται απαραίτητες. Θα συνεργαστώ με τους συναδέλφους. Ελπίζω ότι αυτή η πρόταση θα προχωρήσει και θα μας βοηθήσει στην ε, ενιαία αγορά. Ευχαριστώ κύριο Μέτσαρος. Ε, θέλετε, ευθύνουμε σε εσά. Θέλετε να σχολιάσετε. Όχι, δεν νομίζω λέει ο εισηγητής, δεν χρειάζεται τώρα. Μπορούμε να συζητήσουμε αργότερα, αλλά ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις τη, κυρία Τέιλορ. Και σα εύχομαι, λέει η Πρόεδρος, κάθε επιτυχία για την περαιτέρω συνεργασία, ε, ε σας και προχωρούμε στην, στο σημείο 6 εισηγητής συντάκτη ο κ. Σόμπρο συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωση και της Ρωσική Ομοσπονδία για τις πρόδρομε ουσίε των ναρκωτικών. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, αρχικά θέλω να πω ότι ευχαριστώ ιδιαίτερα τη Γραμματεία και την νομική υπηρεσία της Επιτροπής για την ε, συνεργασία και στην προετοιμασία της γνωμοδότησης. Είναι ένα πολύ ε, ιδιαίτερο θέμα, προφανές θα έλεγα, σήμερα. Αναφέρομαι στη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Είναι πολύ σημαντικό, σημαντική συμφωνία που περιέχει σημαντικά θέματα όσον αφορά την ασφάλεια και την αντιμετώπιση αρνητικών φαινομένων που έχουν σχέση με την ε, παραγωγή συνθετικών ναρκωτικών. Από ό,τι ξέρουμε από αξιόπιστες πηγές η αγορά ναρκωτικών αναπτύσσεται συνέχεια. Τώρα οι οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις ε, εστιάζουν την παραγωγή τους ε, και τις παράνομες δραστηριότητες τους, δηλαδή μεγάλης κλίμακας λαθρεμπόριων ναρκωτικών και εστιάζονται στην, ε, στα συν, συνθετικά ναρκωτικά. Τα ναρκωτικά ξεκαλωθούν και αποτελούν ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τελευταία πέντε χρόνια όμως έχουμε δει μια θετική εξέλιξη, δηλαδή η κατανάλωση ε, παραδοσιακών ναρκωτικών όπως ηρωίνης και κοκαίνης έχει κατά ένα ποσοστό μειωθεί. Αυτό ε, βεβαίως ε, είχε ως αποτέλεσμα να αναπτυχθεί ιδιαίτερα η παραγωγή, κυκλοφορία και εμπορία συνθετικών ναρκωτικών με εξαιρετικά, αρνητικά, με επιπτώσεις επειδή είναι δημοφιλή αυτά τα ναρκωτικά, οι εγκληματικές οργανώσεις τα προβάλλουν ακόμα περισσότερο και αυξάνουν την διαθεσιμότητά τους μεταξύ ορισμένων ομάδων και γι' αυτό θα πρέπει να αναλάβουμε δράση να μειώσουμε πρόσβαση στα πρωτογενή υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται σε αυτές τις εξαιρετικά επικίνδυνες ουσίες. Τα στατιστικά μας στοιχεία δείχνουν ότι η πλειοψηφία των παραγωμένων ναρκωτικών αυτών και τα συστατικά τους εστιάζονται στην επικράτεια της Σοβιετικής Ένωσης, της ε, Ρωσίας, της ε, Ομοσπονδίας Ρωσικό, της Ρωσίας. Και Στο παρελθόν οι προσπάθειές μας επικεντρώνονταν στην, ε, στον περιορισμό της πρόσβασης των πρώτων υλών. Τώρα, έχουμε διαπιστώσει ότι ένα μεγάλο μέρος ε, των πρόδρομων ε, ουσιών κυκλοφορεί στη Ρωσική Ομοσπονδία. Γι' αυτό συμφέρον μας είναι να συντάξουμε μία συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσικής Ομοσπονδίας για την καταπολέμηση αυτής της παράνομης ε, εμπορίας. Γι' αυτό ακριβώς συντάχθηκε αυτή η συμφωνία. Η συμφωνία αυτή εξασφαλίζει επίσης ε, και την προστασία προσωπικών δεδομένων ατόμων που ενδέχεται να σιγούν, να ε, περιληφθούν στις διατάξεις ε, αυτής ε, της συμφωνίας. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά του δεδομένα δεν θα θυγούν, δεν θα παραβιεστούν, ενώ ταυτόχρονα θα εφαρμόζονται πλήρως οι διατάξεις συμφωνίας. Γι' αυτό συστήνουμε στην Επιτροπή να επικυρώσει την τη συμφωνία αυτή, την ολοκλήρωση αυτή τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσική Ομοσπονδία για τι πρόδρομε ουσίε. Η πρόεδρο. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω να θέλει κανείς να λάβει το λόγο. Θέλω να αποσαφηνίσω, λέει η Πρόεδρος, ότι εδώ δεν έχουν υποβληθεί τροπολογίες και γι' αυτό μπορούμε να ψηφίσουμε αμέσως. στη συνεδρίασή μας δηλαδή. Προ... Προχωρούμε στο στην, στον κύριο Μέζαρος με το σημείο 7. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είχαμε συζήτηση πάνω στο θέμα αυτό στην Επιτροπή και θα ήθελα να συνοψίσω και να σα δώσω μια βασική σύσταση πάνω στο θέμα αυτό. Πρόκειται η απόφαση του Συμβουλίου περί εξουδοτήσεω των κρατών μελών που είναι συμβαλόμενη μέρη τη Σύμβαση τη Βιέννη σχετικά με την αστική ευθύνη ω προ τι πυρηνικέ ζημίε τη 21η Μαου του 1953, η πρώτη τη λεγόμενη Σύμβαση τη Βιέννη. Να κυρώσουν το πρωτόκολλο περί τροποποίησεω τη εν λόγω σύμβαση ή να προσχωρήσουν σε αυτό προ το συμφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι ο στόχο τη πρόταση αυτή, Επιτρέπει τα κράτη-μέλη που είναι συμβαλόμενα μέρη τη σύμβαση τη Βιέννη σχετικά με την αστική ευθύνη ω προ τι πυρηνικέ ζημίε, να ακυρώσουν το πρωτόκολλο περί τη τη ελόγω σύμβασης ή να προσχωρήσουν σε, αυτή, σε αυτό. Η απόφαση του Συμβουλίου απευθύνεται στα κράτη-μέλη που είναι συμβαλόμενη μέρη της Σύμβασης της Βιέννης, Βουλγαρία, Τσεχία, Εστονία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Πολωνία και Σλοβακία. αυτή τη στιγμή. Το διεθνές ε, καθεστώς αστικής ευθύνης ως προς τις πυρηνικές ζημίες ε, ε, διέπεται από δύο συμφωνίες, την σύμβαση του, της Βιέννης με το πρωτόκολλο και τη σύμβαση του Παρισιού του 1960 που τροποποιήθηκε με μια σειρά πρωτοκόλων αργότερα και που συμπληρώθηκε από την σύμβαση των Βρυξελών της 31ης ε, ε, Ιανουαρίου του 1953. Και οι δύο αυτές ε, συμβάσεις συμμερίζονται κάποιες από τις βασικές αρχές. Κάποια από τα κράτη-μέλη είναι συμβαλόμενα μέρη της Σύμβασης του Παρισιού, ενώ άλλα κράτη-μέλη είναι συμβαλόμενα μέρη της Σύμβασης της Βιέννης. Η τροποποίηση της Σύμβασης της Βιέννης περιέχει περιέχουν ε, στοιχεία τα οποία να είναι δυνάμει ωφέλιμα για τα θύματα ε, πυρηνικών ζημιών. Αύξηση δηλαδή ε, της ευθύνης και, και γι' αυτό είναι ωφέλιμες για την αποζημίωση των θυμάτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρωτόκολλο που υιοθετήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 1997 υπό την αιγίδα της ε, Διεθνούς ε, Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας ε, περιλαμβάνει ρήτρε σχετικά με τη δικαιοδοσία και την αναγνώριση και επιβολή και εφαρμογή αποφάσεων και Αυτά είναι πτυχές που συμπεριλαμβάνονται στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα στον κανονισμό Βρυξέλλες 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα στι διατάξει αυτέ του πρωτοκόλου και τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να είναι συμβαλόμενοι μέρη του πρωτοκόλλου όσον αφορά τι συγκεκριμένε ε, ρήτρε. Το Συμβούλιο στην απόφαση του προτείνει ε, ε να ε, επικυρώσει τις αποφάσεις του πρωτοκόλου στο όνομα των κρατών μελών. Και Όσον αφορά τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, η απόφαση του Συμβουλίου ζητά ε, συνένεση του ε, Κοινοβουλίου λόγω της αμοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων. Η δική μου σύσταση είναι η εξής. Στηρίζω απόλυτα την πρόταση και συστήνω το Κοινοβούλιο να δώσει τη συνένεσή του. Η διαδικασία αυτή θα επιτρέπει στους συμβαλόμενους ε, της Σύμβασης ε, της Βιέννης ε, να συνάψουν το πρωτοκόλλο του 1900, να προσυπογράψουν το πρωτοκόλλο του 1953. Ίσως να είναι θετικό στο μέλλον να εξεταστεί η δυνατότητα να έχουμε ε, στην ε, Ένωση ενία προσέγγιση όσον αφορά την αστική ευθύνη ως προς τις πυρηνικές ζημιές. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρο. Δεν βλέπω να ζητά κανείς το λόγο. 3 Μαΐου το μεσημέρι είναι η προθεσμία για την υποβολή ε, τροπολογιών και φτάνουμε έτσι στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το υπαριθμόν 8. Ο κύριο Στόγιανοφ είναι ε, συντάκτη τη γνωμοδότηση ε, για το πρόγραμμα τη Ένωση για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα τη χρηματοοικονομικής αναφορά και του λογιστικού ελέγχου κατά την περίοδο 2014 2020. Παρακαλώ κύριε Στογιανόφ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόκειται εδώ για το ότι στοχεύουμε σε μια συμφωνία με το Συμβούλιο για μια νομοθετική πράξη, πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία αφορά την χρηματοδότηση τριών ιδρυμάτων μέσα ε, στο πλαίσιο των, ε, της παρουσίασης των τελικών ισολογισμών. Είναι ένα σύντομο έγγραφο σύντομο και ε, για την επόμενη προγραμματική περίοδο αυτές, αυτά τα τρία ιδρύματα, οι υπηρεσίες πρέπει να χρηματοδοτηθούν για να μην διακοπεί η λειτουργία τους και να μπορούν να επιτελέσουν το έργο τους. Όσον αφορά την παρουσίαση προτύπων, ε, νομικών, νομικών προτύπων, και η βασική ιδέα είναι η δημιουργία ενιαίων νομικών προτύπων σε διεθνές επίπεδο. Στις προ... προηγούμενες ακροάσεις είχα πει ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε και πολλά σε αυτό το θέμα. Έχω μία τροπολογία προτείνει, πρόκειται για τις πράξεις κατεξουσιοδότηση που προβλέπονται στη δική μας νομοθεσία Έχω επίσης, ήθελα να παρατείνω την προθεσμία τροπολογιών και να δώσω τη δυνατότητα στο Συμβούλιο να εγκρίνει τις πράξεις κατ' εξουσιοδότηση από πλευράς κομισιών. Συζήτησα με εμπειρογνώμονες του κλάδου και με... μου εξήγησαν γιατί αναφέρονται σε αυτό το κατάλογο, αυτά τα πρόσωπα και που ζητούν αυτά τα κονδύλια. Αυτές οι υπηρεσίες, αυτά τα ιδρύματα είναι πολύ σημαντικά σε διεθνές επίπεδο ε, και ε, πρέπει ε, θέλουμε να ελαφρύνουμε το λογιστικό έλεγχο και τις χρηματοοικονομικές αναφορές που γίνονται από πλευράς ιδρυμάτων. Αυτό είναι υποχρεωτικό, είναι υποχρεωτική η επιβολή των λογιστικών στοιχείων και των, ε, του έτους. Οι οργανώσεις, ιδρύματα, οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην πρόταση νομοθετικού περιεχομένου χρηματοδοτούνταν μέχρι τώρα αποκλειστικά από τα κράτη-μέλη. Και τα κράτη-μέλη ήταν οι ιδρυτές αυτών των φορέων. Στο, στην τελευταία προγραμματική περίοδο είχε διακοπεί αυτή η χρηματοδότηση η οποία τώρα θα πρέπει να καλυφθεί από μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχα πει ότι θα εκδώσουμε μία σύσταση σε, αυτά τα, σε αυτούς τους φορείς ε, επί τη βάση της κοινοτικής χρωματοδότησης. Και η σύσταση θα λέει ότι θα υπόκεινται στο λογιστικό έλεγχο και σε όλους τους ελέγχους που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θα προτείνω μία τροπολογία οι τροπολογίες θα έχουν το χαρακτήρα σύστασης και ο στόχος μου είναι η εδραίωση της επιθαρχίας και της διαφάνειας. Μία, ένας τέτοιος φορέας, το, το εκτελεί ήδη αυτό, είναι για τις άλλες δύο περισσότερο που ισχύει αυτή η χρηματοδότηση, η χρηματοοικονομική αναφορά. Η πρόεδρος, ευχαριστώ. Άλλες, ε, άλλος επιθυμεί να παρέμβει προθεσμία. Ε, τροπολογιών είναι... Α, ...8 Μαΐου είναι η λήξη της προθεσμίας τροπολογιών. Ολοκληρώσαμε και το 8, το θέμα 8 και προχωρούμε στο 9. Καθεστώς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος. Ενδιάμεση έκθεση. Κυρία. Α, και εγώ θα δώσω το λόγο στον εαυτό μου. Καταρχάς, λυπάμαι που λείπουν οι σκιώδεις εισηγητέ. Οι εισηγήτριε, η κυρία Φροτάν και ο κύριος Κάντης Πασκουάλ και τους ευχαριστώ για τις τροπολογίες τους και μπορώ να πω ότι οι τοπολογίες αυτές είναι πολύ χρήσιμες ε, και χωρίς κανένα πρόβλημα θα μπορέσω να τις ενσωματώσω στην έκθεσή μου και σε συνεργασία με την Επιτροπή Πολιτισμού και την αρμόδια συγγήτρια, την κυρία Χίρς, Έχουμε συνεργαστεί επικοδομητικά και εκείνη έχει υποβάλει τροπολογίε που μπορώ να ενσωματώσω έτσι ώστε να επιτύχουμε τους καλύτερους συμβιβασμούς. Θα αναφερθώ καταρχάς στις τροπολογίες του κυρίου Γκράντε Πασκουάλ και είναι πολύ θετικό αυτό το οποίο προτείνει σε σχέση με την, τον ορισμό των, ε, της της αξίας, της περιουσιακής αξίας για την ε, πρόσταση και την επιβολή προστιθέμενες αξίες στη λειτουργία, στο καθεστώς και τονίζω και την τροπολογία του 12 η οποία ζητάει περισσότερη διαφάνεια. Συμφωνώ απολύτως. Ε, θα πρέπει ίσως να συζητήσουμε περαιτέρω την διεύρυνση του καταλόγου με τα συν και τα πλήν στις τροπολογίες και δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνάμε το φορολογικό καθεστώς όπου υπάρχουν θετικά και αρνητικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να αναλύσουμε με μεγάλη προσοχή. Επίσης συμφωνούμε στη, στο διασυνοριακή πτυχή, η οποία θα πρέπει να είναι παρούσα, δηλαδή πρέπει να είναι σαφέστατο ότι το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα ε, θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον δύο κράτη-μέλη. Ε, πρέπει να συζητήσουμε ορισμένες άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί όσον αφορά τις ε, διαφορές που προκύπτουν από τα μέλη των οικογενειών. Εδώ αυτές τις τοπολογίες, αυτό το περιεχόμενο πρέπει να τις συζητήσουμε περαιτέρω και να τις διατυπώσουμε καλύτερα. Αυτή είναι η επιστημία μου. Επίσης δεν καταλαβαίνω απόλυτα το ζήτημα της διαγραφής των άρθρων για την φορολόγηση. Ε, τι ακριβώς εννοεί ο συντάκτης. Όσον αφορά τις απολογίες της κυρία Τάιν, η μείωση των οικονομικών δραστηριοτήτων από 10 σε 5% καθαρού ετήσιου κύκλου εργασιών είναι καλή ιδέα, μπορώ να τη δεχθώ και άλλο ένα σημαντικό στοιχείο, και εδώ έχω μεγάλες επιφυλάξεις, είναι όσον αφορά τους απασχολούμενους. Εδώ. Δεν θέλω να δεχτώ την αρχική διατύπωση της Κομισιόν για τους επίτιμους, επίτιμους, τις επίτιμες θέσεις ε, δεν καταλαβαίνω γιατί η Κομισιόν έχει παρεμβάλει αυτή την πρόταση στην πρότασή της. Ε, διότι φαίνεται ότι σε αυτό τον τομέα απασχολούνται πολύ επίτιμοι. Και ε, αυτές ήταν οι βασικές μου παρατηρήσεις και προσβλέπω με μεγάλη χαρά την συνεργασία μας και πιστεύω ότι στα θέματα που ακόμα υπάρχει διαφορετική αντίληψη να μπορέσουμε τελικά να ε, συγκλίνουμε. Και δίνω αμέσως το λόγο στο σκιώδη εισηγητή κύριο Λουίς Ντεγκράντες Πασκουάλ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη, έφτασα τρέχοντας και καθυστερημένος αυτή είναι η μοίρα μας εδώ στο Κοινοβούλιο. Άκουσα όμως τα τελευταία σας τουλάχιστον λόγια και θα ξεκινήσω από αυτά. Συμφωνώ βέβαια. Είναι αλήθεια ότι έχω υποβάλει 14 τροπολογίες, αλλά εξ αρχής θέλω να δηλώσω ότι ε, το πνεύμα τους είναι συμβιβαστικό. Θέλω να συμβιβάσω την άποψη των σκιωδών συγκοητών, άλλων συναδέλφων που έχουν υποβάλει ε, προτάσεις ε, τροπολογίας και πιστεύω ότι μπορούμε να συγκλίνουμε διότι δεν έχουμε μεγάλες συγκρούσεις μεταξύ μας. Να σας αναφερθώ στις δικές μου τροπολογίες, αλλά να πω ότι από τις τρεις ε, τροπολογίες της συγκήτριας, εκτός από μία που μου δημιουργεί δισταχμούς, οι υπόλοιπε μας βρίσκουν σύμφωνος. Είμαστε υπέρ ε, της τροπολογίας του κ. Μασίπ επίσης. Σε ό,τι αφορά την κυρία Τέιν που έχει υποβάλει έξι τροπολογίε, μπορώ να πω ότι πέντε με βρίσκουν σύμφωνο. Την έκτη θα τη συζητήσουμε. Οπότε βλέπετε, δεν έχουμε μεγάλη απόκληση. Αυτό που εγώ πρέπει να σας εξηγήσω όμως είναι το σκεπτικό πίσω από τις δικές μου τροπολογίες. Καταρχήν τροπολογία 1. Άρθρο 2 ορισμοί. Ε, θέλουμε να προσθέσουμε ε, τον όρο ε, οικονομική κοινωνική αξία, όχι σκέτα, σκέτο αξία. Οι τροπολογίες 3 και 4 ε, που αφορούν το σκοπό των Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων Προσθέτουμε μεταξύ των σκοπών και την ε, συνδρομή στα θύματα της τρομοκρατίας και, της, ε, και πράξεων βίας ε, και επίσης την προώθηση του θρησκευτικού διαλόγου. Νομίζουμε ότι και τα δύο αυτά ζητήματα είναι επίκαιρα και τα οποία ως τώρα εξαιρούντο του δεν καλύπτονταν τουλάχιστον από τον κατάλογο ε, των ε, σκοπών τα οποία, τους οποίους θα έπρεπε να έχει ή θα μπορούσε να έχει ένα ε, ίδρυμα, ευρωπαϊκό ίδρυμα. Τροπολογία 7. Η, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα θα πρέπει να έχει δραστηριότητες σε παραπάνω του ενός κράτη-μέλη. Τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα. Ε, λέει τη στιγμή της καταχώρησης. Θα το διέγραφα, γιατί θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Η υποχρέωση θα πρέπει να είναι μόνιμη, γιατί αλλιώς μπορεί να εγγραφεί, να καταχωρηθεί ε, με δραστηριότητα σε πολλά κρατημέλη και μετά να το τροποποιήσει, να τροποποιήσει το καταστατικό του το Ίδρυμα. η διαγραφή έχει σχέση με το ότι σίγουρα θα πρέπει στην εγγραφή, στην καταχώρηση ε, το Ίδρυμα να ε, δηλώνει ότι έχει δραστηριότητα σε περισσότερα τρόνους κάτι μελη αλλά αυτό θα πρέπει να είναι μόνιμο. Αν συμφωνούμε με αυτό, δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα με τη διαγραφή της συγκεκριμένη φράσης. Τροπολογία 10. Τροποποιούμε το κείμενο, το τελευταίο κομμάτι, λέμε υπό την προπόθεση ότι δεν θα απαγορεύεται από το ε, καταστατικό και δεν θα είναι αντίθετη με την ε, βούληση του ιδρυτή. Μιλάμε για την ε, δημιουργία ιδρύματος ε, μέσω μετατροπής ε, μια, ενός δημόσιου φορέα. Τροπολογία 12. Κατάλογος των εγγράφων ε, και δικαιολογητικών που θα πρέπει να παράσχονται, καθώς επίσης και των στοιχείων, όνομα, όνομα επώνυμο, η διεύθυνση των ε, ιδρυτών και, και προσθέτουμε και την ε, ε, έδρα των νομικών προσώπων. Για τα νομικά πρόσωπα ή η διεύθυνσή του, η ταχυδρομική του διεύθυνση δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η σημασία είναι που έχουν την καταστατική του έδρα. Νομίζω ότι και αυτή η πρόταση δεν θα πρέπει να βρει αντίθετους. Τροπολογίες 13 και 15. Δεν θέλουμε να εξαιρεθούν από τα ωφέλη ε, ορισμένα άτομα τα οποία ε, έχουν σχέση με τη διαχείριση των ιδρυμάτων και οι οικογένειε του. Ε, τα ευρωπαϊκά ιδρύματα ε, είναι, έχουν ε, μη κερδοσκοπικό σκοπό. δεν θα πρέπει να τα συγχαίουμε με την εμπειρία των οικογενειακών ιδρυμάτων που στην Ισπανία τουλάχιστον έχουν πολύ καλή εμπειρία και με αυτά. υπάρχουν τέτοιου ιδρύματα για να εξασφαλιστεί η σωστή διαχείριση της περιουσίας συγκεκριμένων οικογενειών, ε, για παράδειγμα μιας ε, συλλογής ε, πινάκων ζωγραφικής ή κάποιας ακίνητης περιουσίας επίπλων κλπ. κλπ. τέτοιου είδους συλλογές δορίζονται στο κράτος αλλά την χάνουν διαχείρισης από ιδρύματα οικογενειακά. Δεν θέλουμε λοιπόν να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε κάτι το οποίο δεν είναι δυνατό να περιοριστεί. Πρόκειται για διαφανείς διαδικασίες που ε, γίνονται για λόγους νόμιμους και θεμητούς. Μετά, η 15 έχει σχέση με το εργασιακό καθεστώς. Ε, εγώ είχα εκφράσει κάποιες αντιρρήσεις και ε, ε, δισταγμούς για το θέμα των εθελοντών. Νομίζω ότι είναι υπερβολικό να δεχόμαστε ότι μπορούν να συμμετάσχουν. Μπορούν να ενημερώνονται, αλλά όχι και να συμμετάσχουν. 41 για το άρθρο 44. Ε, συγγνώμη, 21 για το άρθρο 44 τώρα. Ε, προσθέτουμε το κείμενο με έδρα στο ίδιο κράτος μέλος το οποίο είναι εγγεγραμμένο το Ίδρυμα. Ο στόχος είναι ε, η περιουσία να μπορεί να ε, μεταφερθεί σε άλλο φορέα ή ε, κρατική οντότητα που θα έχει έδρα στο ίδιο κράτος μέλος. Γιατί ασφαλώς το κάθε κράτος μέλος θα έχει τις ε, θεμητές του απαιτήσει σε τέτοιου είδους ε, περιπτώσεις. Τέλος, τροπολογίες 22, 23 και 24. Προσπαθούμε να διαγράψουμε τα άρθρα σχετικά με τη φορολόγηση. σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη με τα οποία ήρθαμε σε επαφή ε, κατά κανόνα συμφωνούν. Το Υπουργείο Οικονομικών στην Ισπανία το, το ανέφερε ρητά άλλωστε. Ανεξαρτήτως δογμάτων και ιδεολογιών, είναι σημαντικό να δούμε ότι ε, σε αυτό το θέμα ε, συμφωνούν ε, όλοι. Τώρα, η... επαναλαμβάνω ότι πρόθεσή μου είναι να είμαι συμβιβαστικός, επικοδομητικός. θέλω να βρούμε συμβιβασμό με την εισηγήτρια, με τους και εισηγητές. Η εισηγήτρια των φιλελευθέρων έχει υποβάλει ενδιαφέρουσε τροπολογίες. Η τροπολογία του Κορμασίφ είναι επίσης ενδιαφέρουσα και αποδεκτή. Το δικό μου πνεύμα είναι αυτό, το συμβιβαστικό επικοδομητικό πνεύμα. Και έχω την εντύπωση, αν να μην πω βεβαιότητα, ότι δεν μας χωρίζει χάος. Νομίζω θα βρούμε μια μέση λύση. Αυτή θα είναι η δική μου πρόθεση και προσπάθεια. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις ε, παρατηρήσεις σας, διότι απαντήσατε σε διάφορα ερωτήματα και δίνω το λόγο στην κυρία Τάιν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ σύντομα στις τροπολογίες. Κατ' εξαίρεση, να αναφερθώ στην τροπολογία ενα του συναδέλφου Τεκράντες. Δεν ξέρω αν αυτό σχετίζεται με την ε, γερμανική αγγλική μετάφραση, αλλά ε, ο γερμανικός όρος δεν συμπεριλαμβάνει μόνο τους υλικούς σπόρους, ε, συμπεριλαμβάνει και ε, άειλους, ε, πνευματικούς κλπ. Δεν θα συμφωνούσα λοιπόν με διαφορετική ορολογία στα γερμανικά. Επίσης όσον αφορά την συναπόφαση, συμφωνώ με το ΕΛΚ το θέμα εδώ είναι η άμυστη. Αν ε, εγώ έχω μία άμυστη θέση και κάτι δεν μου αρέσει, εάν θεωρώ ότι από τον εργοδότη μου εντός εισαγωγικών ε, δεν ε, λαμβάνω την σωστή αντιμετώπιση, τότε μπορώ να αποσυρθώ. και έτσι να ασκήσω πίεση στον, ε, στον, υπεύθυνο, ενώ ένας ε, εργαζόμενος δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Είναι λοιπόν πολύ διαφορετική η κατάσταση ανάμεσα στους ε, κανονικούς εργαζομένους ε, και τους άμυστους. Προέρχομαι από χώρα που που εκτιμά ιδιαίτερα το θέμα της συναπόφασης. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι το συγκεκριμένο θέμα αυτό θα περνούσε από την Ολομέλεια και να, εξηγήσω την τροπολογία μου υπαριθμών 17, όπου λέω ότι η η γνωμοδότηση δημοσιοποιείται σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους μέλους. Ε, δεν καταφέραμε να πετύχουμε συμφωνία στο θέμα αυτό και γι' αυτό δεν ξέρω καν αν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την νομοθετική διαδικασία, αλλά ε, υποθέτω ότι θα συνεχίσουν να ισχύουν οι νομοθετικές διατάξεις που ίσχυαν μέχρι τώρα και στην ε, Γερμανία αν έχουμε μια, 400, ε, μια ε, γνωμοδότηση 400-500 σελίδων σύμφωνα με τον συγκεκριμένο κανόνα θα πρέπει να κοινοποιείται όλοι. Οι περισσότερες πληροφορίες όμως δεν προορίζονται για το ευρύ Παρακαλώ λοιπόν να λάβουμε υπόψη τις ισχύουσε διατάξει ε, στο κάθε κράτος μέλος. Τα περισσότερα κράτη-μέλη δεν γνωρίζουν καν ε, αυτήν την γνωμοδότηση για τον έλεγχο των λογαριασμών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ. Και τους δύο εισηγητές για τις ε, τις παρατηρήσεις και τα σχόλια τους. Όσον αφορά τώρα τις άμυστες ή εθελοντικές θέσει, θα ήθελα να ακούσω την άποψη της Κομισιόν, τον κύριο ε, Βέρμαν, να μας βοηθήσει λίγο, να μας ενημερώσει λίγο ποια είναι η κατάσταση και ποια είναι τα στοιχεία στα οποία μπορούμε να βασιστούμε. Πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό, διότι πιστεύω ότι η Κομισιόν ε, πριν ε, παρουσιάσει την πρότασή της την έχει πολύ καλά μελετήσει. Είναι κάποιος εκπρόσωπος της Κομισιόν εδώ. Πείτε. Yeah, thank you. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για θέσεις επί, επίτιμες, εννοείται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έτσι δεν είναι επίτιμα μέλη. Ε, στα γερμανικά λέγεται Ehrenamtlich, που μπορεί να είναι και εθελοντές και άμυστοι. Ε, και η κυρία Τάιν αναφέρεται και στη συναπόφαση και τη συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια. Αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια αντιπρόθεση η σας να συμπεριλάβετε κι εσείς αυτού του τύπου τους εργαζόμενους ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την επεξήγησή σας. Για να είμαστε σαφείς για τους εθελοντές. Εθελοντές στα ιδρύματα είναι γενικά πολύ σημαντικοί εργαζόμενοι, διότι δουλεύουν μέσα στα ιδρύματα, για τα ιδρύματα. Εάν κοιτάξουμε το νομικό πλαίσιο στα κράτη-μέλη, είναι σαφές ότι δεν υπάρχει το αντίστοιχο νομικό πλαίσιο σε όλα τα κράτη-μέλη για τους ε, εθελοντές. Έχοντας υπόψη ότι θέλαμε να προτείνουμε ε, ένα... Ε, ένα ίδρυμα το οποίο είναι πολύ προοδευτικό και το οποίο λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα όλων όσων ασχολούνται με το έργο του θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη και το καθεστώς των θεσελοντών που συμμετέχουν στις εργασίες των Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων. Αυτό που βλέπουμε στο Συμβούλιο αυτή τη στιγμή είναι ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη έχουν μεγάλες επιφυλάξεις στο να δημιουργηθεί ένα ειδικό πλαίσιο για εθελοντές εργαζόμενους και οι περισσότεροι θα ήθελαν να τηρήσουν το εθνικό του σύστημα, εάν υπάρχει, εάν και εφόσον υπάρχει. Αυτό μπορώ να σας πω εγώ από τη στιγμή για τους volunteers, τους εθελοντές. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ, η κυρία Τάιν, όσον αφορά τους άλλους. Ίσως υπάρχει μια παρανόηση και πρέπει να την αποφύγουμε. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να προβλεφθεί αυτό στην πρόταση και να ενημερώνονται ε, θελοντές ε, για, τις, ε, για το έργο ούτε έχω και καμία αντίρρηση να προστατεύονται με το εργασιακό καθεστώς των άλλων. Αυτό για μένα είναι προφανές. Όμως, όταν υποβάλλονται τροπολογίες που λένε ότι οι εθελοντές, οι θα πρέπει να βρίσκονται στην ίδια μοίρα ε, όπως και οι άμυστοι και ότι θα πρέπει να καλυφθούν από τα δικαιώματα συναπόφασης. Τότε εγώ το ερμηνεύω αυτό ως εξή ότι σε όλες τις συνεδριάς του Διοικητικού Συμβουλίου θα εκπροσωπούνται για να μπορούν να επιτελέσουν ε, και με δικαίωμα ψήφου μάλιστα ε, το, το, τη διαδικασία της συναπόφασης. Τώρα, εάν δεν υπάρχει κάποιος άμυστος ή εθελοντής που συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, τότε θα μπορούσε αυτό να ερμηνευτεί ότι του αφαιρείται το δικαίωμα να συμμετάσχει στη διαδικασία συναπόφασης. Τώρα, δικαίωμα προστασία στην εργασία, αυτό είναι προφανές. Sí, ο κ. Πασκουάλ. Η Κομισιόν δεν μας διευκρίνησε πολλά. Η παρέμβαση της ηγήτρας όμως κυρία Στάι, Τάιν με διευκρίνησε πολύ περισσότερα. Συμφωνώ. Ο σκοπός δεν είναι να αρνηθούμε στους εργαζόμενους στρίκτου σένσου την συμμετοχή τους. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι κάθε χώρα έχει διαφορετικό καθεστώς που διέπει τους εθελοντές. Στην Ισπανία τους δίνουμε όλο και περισσότερες δυνατότητες συμμετοχής, αλλά ε, άλλο όμως είναι αυτό που προτείνει η Κομισιόν, ότι οι εθελοντές θα συμμετέχουν υποχρεωτικά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος και θα μπορούν έτσι να ε, επηρεάζουν την πολιτική του. Με αυτό διαφωνώ. Δεν είναι δυνατόν να τους εξισώνουμε με τους ε, εργαζόμενους του Ιδρύματος και να τους δώσουμε φωνή και ψήφο στα διοικητικά συμβούλια. Η Κομισιόν νομίζω ότι είναι υπερβολική στις απαιτήσει Εμείς θέλουμε να μειώσουμε λίγο αυτό το πεδίο το οποίο έχουν, έχει προβλέψει η Κομισιόν. Συζητήτρια, θέλω να παρατηρήσω το εξής. Στην τροπολογία σας εκφράζεται την επισημία οι θέσει αυτές να έχουν το καθεστώς που, λέει ότι έχουν το καθεστώς του παρατηρητή να διαγραφεί. Ως αυτό υπερβαίνει τους στόχους. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί που απασχολούνται θελοντικά ή αμυστοί που υπόκεινται σε διαφορετικές εθνικές ρυθμίσεις και ε, νομοθεσίες, σε αυτούς θα πρέπει να τους διαχωρίσουμε από τα, αυτούς που συμμετέχουν και έχουν δικαιώματα στην απόφαση στα διοικητικά συμβούλια. Εμέ με απασχολεί πάντοτε το θέμα της εθελοντικής εκπροσώπησης και θέλω να υπάρχει συνοχή μεταξύ αυτού του θέματος των Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων, του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος και άλλων Ιδρυμάτων όπου υπάρχει το ίδιο εργασιακό καθεστώς. Θα έλεγα λοιπόν στους εισηγητές να εξετάσουμε αυτό το θέμα εις βάθος με, και να οργανώσουμε μία συνάντηση με τους σκιώδεις εισηγητής για να διευκρινίσουμε αυτό το θέμα, για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μία συμφωνία. Δόξα το Θεό, από ό,τι φαίνεται έχουμε τη δυνατότητα καλών συμβιβασμών. Και η 30 Μαΐου είναι η προθεσμία ε, για να ψηφίσουμε αυτό το θέμα και μέχρι τότε έχουμε καιρό να επιτύχουμε μια συμφωνία, μια σύγκληση απόψεων. Και έτσι ολοκληρώσαμε την ημερήσια διάταξη. Για το πρωί, το απόγευμα θα συνεχίσουμε με τον ε, δομημένο διάλογο με την ε, αντιπρόσωπο της Επιτροπής, την κυρία Ρέντινγκ και ο κύριος Λέιν θα είναι πάλι εδώ, θα αναλάβει ο πρόεδρος ε, την Προεδρία της Επιτροπής και ούτω πώς ε, ολοκληρώνω την πρωινή μας συνεδρίαση.